Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask... Χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. And we'll be able to begin our... Αρχίζουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. I open the Regi meeting for today. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής. Έγκριση σήμερα διάταξη είναι το πρώτο θέμα. Έχω να σας κάνω ανακοινώσεις για την ημερήσια διαταξή τη σημερινή. Την Πέμπτη στο Στρασβούργο η διάσκεψη των Προεδρών αποφάσισε να αναβάλει την απόφαση σχετικά με το ποια επιτροπή θα είναι αρμόδια για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για το πρόγραμμα στήριξης διαστατικών μεταρρυθμίσεων. Αναβλήθηκε λοιπόν η απόφαση αυτή. Συνεπώς, η ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο κύριο Ντομπρόφσκι που είχαμε ως σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη στο σχέδιο, αναβάλλεται και αυτή μοιραία ε, για ευθετότερο χρόνο. Ενημερώθηκαν οι βουλευτές ε, την περασμένη Παρασκευή και αυτή είναι η αλλαγή στην ημερήσια διάταξή μας για τη σημερινή συνεδρίαση. Ε, λοιπόν, όταν θα λάβουμε την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με το ποια επιτροπή θα αναλάβει λοιπόν, θα ε, σας προτείνουμε μάλλον μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής το Μάιο ή αρχές Ιουνίου. Θα δούμε. Μόλις αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων και μετά θα αποφασίσουμε κι εμείς. Ε, Ούτω λοιπόν έχει αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Προτείνετε τίποτα, έχετε να ρωτήσετε. Κύριε Βανίστε Ρόι, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Προτείνω να αρχίσουν αμέσω μετά οι συντονιστέ στι 4.30 δηλαδή, νωρίτερα. Ναι, βεβαίω, να μην χάσουμε χρόνο. να Αρχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών αμέσω μετά την ολοκλήρωση τη ε, σημερινή ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν δεν έχετε άλλες ερωτήσει για την σε διάταξη. Θεωρούμε ότι εγκρίνεται με την αλλαγή αυτή. Δύο ανακοινώσει έχω επιπλέον του Πρόεδρου. Με τη Πρόεδρου καλύτερα πρώτη. Έχει να κάνει με την απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων για το θέμα αυτό, για το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ήταν η πρώτη που σας έκανα. Η δεύτερη και πάλι ενημερωτικά. Η επόμενη συνεδρίαση της διάσκεψης ε, θα λάβει χώρα στις 4 Μαΐου και μόνο ε, μετά τη συνεδρία θα γνωρίζουμε αν θα είμαστε αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Ρέγγι ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης αν ισχύει αυτό, θα ζητήσω από την Γραμματεία να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση που θα αφιερωθεί ακριβώ στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντομπρόφσκη, αρμόδιο επίτροπο και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ημερομηνίε. Θα τι μάθουμε αργότερα και προσβλέπω και ελπίζω να έχω την υποστήριξη των συντονιστών σε αυτό. Δεύτερη ανακοίνωση. Αντιπροσωπεία στη Μαρτινίκα. Όπως γνωρίζετε, στείλαμε και την προσωπία ε, τη εβδομάδα μετά το Καθολικό Πάσχα. Επικεφαλής ήταν ο κύριος Τσέλερ και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μας κάνει μια σύντομη ενημέρωση έκθεση των πεπραγμένων εκεί της ε, προσωπία μας στην Μαρτινίκα και τι δουλειά κάνατε. Ναι. Ε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, η Μαρτινίκα, όπως και άλλες περιφέρειες, εκτός, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Υπήρου και ανήκει στις λεγόμενες ε, άκρος απομακρυσμένες περιφέρειες ή εξόχως απομακρυσμένες που έχουν ιδιαίτερη ε, θέση στο πλαίσιο των συνθήκων και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνθήκη της Λισαβόνας επίσης προβλέπονται ειδικέ εντάξει. Ανήκει στη Γαλλία η Μαρτινίκη βεβαίω, αλλά ε, βρίσκεται στην Καραϊβική. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μοσκούρ που είχε την ιδέα να επισκεφθούμε τη Μαρτινίκ. Η δική μας επιτροπή είναι αρμόδια για τις περιοχές αυτές, τις ιδιαίτερα απομακρυσμένε, αλλά ε, και μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει πώς ε, θα μπορούμε να τις υποστηρίζουμε. Αν συγκρίνουμε τις διάφορες περιφέρειες μεταξύ τους, έχουν τεράστιες διαφορές προφανώς. Και για να τις καταλάβει κανείς πρέπει να μεταβεί εκεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους, με τους αρμοδίους φορείς και αρχές του τόπου. <clears throat> Έτσι έγινε και στη Μαρτινίκ. Είναι ένα νησί της Καραϊβικής και πριν από τρία χρόνια, γιατί έχουν περάσει τόσα πολλά, είχαμε πάει στην Γαλλική Γουιάννα και ε, εκεί οι αρμόδιοι φορείς μας είπαν ότι η Γαλλική Γουιάννα ως τμήμα της Ευρώπης ε, πλήττεται σφόδρα από τη μετανάστευση, νόμιμη και παράνομη. Ενώ στη Μαρτινίκα, επειδή είναι μεγάλη ανεργία και επειδή δεν υπάρχουν ευκαιρίες για δουλειές, Πολλοί νέοι φεύγουν από το νησί. Άρα υπάρχει και ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα πλέον. Βλέπετε ότι είναι κοντινές περιφέρειες, αλλά αμέσως αμέσως φαίνονται οι τεράστιες διαφορές που επικρατούν και οι διαφορετικές συνθήκες. Το πρόγραμμά μας ήταν πάρα πολύ πυκνό, πάρα πολύ ευρύ, ε, για να δούμε όλα τα προβλήματα, ε, όλα τα ζητήματα και όλες τις δυνατότητες. Ε, που ε, διανοίγονται εκεί. Την πρώτη μέρα επισκεφτήκαμε ένα νέο κτίριο, ένα νοσοκομείο που είναι καινούριο και έχει την ιδιαιτερότητα την εξή. Επειδή είναι σεισμογενή η περιοχή, έπρεπε να είναι αντισυσμικό το κτίριο, πράγμα που καταλαβαίνετε ότι εκτόξευσε και το κόστος και δυσκόλεψε και την κατασκευή ε, του κτίριου, την ανέγερση. Από πλευρά διαστάσεων το νοσοκομείο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κεντρικό νοσοκομείο για όλη την ε, περιφέρεια εκεί. Ωστόσο, και πάλι, αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία που έχουν οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές στη Μαρτινίκα, όπως και στην συνολή Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ευρωπαϊκέ προδιαγραφές και πρότυπα, άρα και γαλλικές, επομένω είναι αφού είναι στη Γαλλία. Ανοίξει η Γαλλική Δημοκρατία. Και αυτό επηρεάζει βεβαίως και την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες περιοχές. Γιατί και στην οικονομία και άλλο θα πρέπει να καταβάλει το ελάχιστο μισθό που ισχύει δια νόμου στη Γαλλία. Ενώ στα κοντινά νησιά γύρω-γύρω επικρατούν άλλες συνθήκες και εργασιακές και στα κοινωνικά και στα διάφορα άλλα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ευρωπαϊκό και το γαλλικό δίκαιο. Πώς λοιπόν θα λυθεί αυτό. Είναι ένα, ένα πρόβλημα. Εάν έρχονται ασθενείς από την Καραϊβική σε αυτό το νοσοκομείο ή ακόμα και από την Αμερικανική Ήπειρο, την Υπηρωτική ε, χώρα πώς θα έχει υπερίθαλψη αυτών των ασθενών. Πρέπει να συναυθούν ε, συμβόλαια και να γίνουν συμφωνίες για να αξιοποιηθεί αυτό το περιφερειακό νοσοκομείο. Πρόκειται να ανοίξει σύντομα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το έργο και θα είναι από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της περιφέρειας εκεί. Επίσης, συζητήσαμε και με αγρότες είναι μέγας ε, κλάδος και της οικονομίας η καλλιέργεια μπανάνας και τα αγροκτήματα είναι μικρομεσαίας ε, έκτασης. 3 με 5 εκτάρια είναι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και η πιο μεγάλη μπορεί να είναι 100. Καλλιεργούν μπανάνα. Ξέρετε ότι αυτή η καλλιέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη έχει πολύ μεγάλη ένταση εργασία. Δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίε για δουλειέ μεν, πλην όμω. Και πάλι οι προδιαγραφές είναι οι ευρωπαϊκές και οι γαλλικές που θα πρέπει να καταβάλλονται αντίστοιχοι μισθοί στον Ισημερινό, στην Κεντρική Αμερική και στην Κολομβία οι μεγάλες εταιρείες μπανάνες δεν έχουν ε, ε, να πληρούν τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, άρα η ανταγωνιστικότητα πέφτει. Αυτό αφορά και τα Κανάρια νησιά που είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες και καλλιεργείται μπανάνα. Σε ό,τι αφορά τι ποσοστώσει δηλαδή και τέτοια ζητήματα και κρατικέ ενισχύσει είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αυτό. Άλλο σημαντικό παράγον είναι η καλλιέργεια του ζαχαροκαλάμου και ε, η επεξεργασία του κάνουν, ε, βγάζουν ζάχαρη και ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Στη Μαρτινίκα ένα πάρα πολύ καλό ρούμι από ζαχαροκάλαμο και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η προστασία του σήματος, ε, του εμπορικού σήματος. Και είπαμε στους συναδέλφους εκεί ότι Βεβαίω, πρέπει να το κάνουν και μπορούν να ασχοληθούν και να επιληφθούν και να το ζητήσουν. Είχαμε επίση συναντήσει με του δημάρχου των διαφόρων εκεί δήμων. Και προηγουμένω, βεβαίω και με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο που είναι και αρμόδιος για τα διαρθρωτικά προγράμματα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Μαρτινίκα έχει επίσης αποφασιστεί πρόσφατα και τώρα μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται. Μέχρι το 2020 είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ τα κονδύλια που τους αναλογούν από τα διαρθρωτικά ταμεία. Κάτι που μας έκανε εντύπωση και μας προξένει έκπληξη είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμαρχη δηλαδή, σχεδόν δεν έχουν ενημέρωση καμία για το ΕΣΠΑ, για το, τα προγράμματα αυτά τα επιχειρησιακά που έχουν αρχίσει και τρέχουν. Δηλαδή είναι ζήτημα επικοινωνίας. Εκείνων που είναι αρμόδιοι επιτόπου, στην περιφέρεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση για τα έργα, θα πρέπει να γνωρίζουν τι ισχύει Και χωράει μεγάλη βελτίωση εκεί. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και οι αυτοδιοικητικοί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να γνωρίζουν και να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και στην εκπόνηση των προγραμμάτων των επιχειρησιακών, αλλά κυρίως και στην εκτέλεση και την υλοποίηση. Δεν γίνονται τα σωστά έργα και τα κατάλληλα κάθε φορά. Είδαμε και εκπροσώπους των οικονομικών, των παραγωγικών τάξεων ιδιαίτερα σε εκείνους που εργάζονται με τα πίεση γεωργικών προϊόντων. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους επιμελητηρίων. Σημαντικός κλάδος της οικονομίας είναι και ο τουρισμός φυσικά στη Μαρτινίκα. Μπορούν να δημιουργηθούν εκεί, να διατηρηθούν και οφείλουν να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Ένα έργο που τελείωσε μόλις με ευρωπαϊκά κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι το εξή. Μέχρι τώρα ε, οι μετακινήσεις γινόντουσαν με γιοταχή ή ε, ατομικά και τώρα δημιουργήθηκε ένα σύστημα συγκοινωνιών δημοσίων από την πρωτεύουσα ε, Fort de France και γύρω από την πρωτεύουσα και μέσα στην πρωτεύουσα αστικές και περιαστικές συγκοινωνίες, πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα. Δεν μας έκρυψαν επίσης ότι Αντιστάθηκαν οι οδηγοί ταξί που δεν θέλησαν ε, να δημιουργηθούν αυτές οι αστικές συγκοινωνίες γιατί θεώρησαν ότι θα επιδίνουν τη δική τους θέση ε, γιατί κάλυπταν και με ιδιωτικά ταξί αυτές τις μεταφορές αλλά νομίζω ότι θα διασκεδαστούν αυτοί οι φόβοι και ανησυχίε του. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί ο κόσμο στο Fort de France και γύρω-γύρω να κυκλοφορεί με τι αστικέ συγκοινωνίε. Και μάλιστα Αυξάνεται και ο πληθυσμός της πρωτεύουσα σε αντίθεση με άλλες ε, πόλεις ε, του νησιού. Με αυτή την αστική συγκοινωνία λοιπόν λεωφορεία δημιουργήθηκε και δική ε, λεωφοριολορίδα και γίνεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία και οι συγκοινωνίες. Σύντομα τώρα για τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις για την ιδιαίτερη κατάσταση στη Μαρτινίκα. Έχουμε γράψει ένα κειμενάκι στο Reggae News, σε αυτό το ενημερωτικό μας δελτίο. Ευχαριστώ τους κύριους Οργάσκη και την κυρία για από τη Γραμματεία. Έχουμε και ένα έγγραφο αγγλικά και γαλλικά, μια περίληψη, έκθεση πεπραγμένων της αντιπροσωπείας εκεί και μπορείτε να ενημερωθείτε για την σύνθεση και της αντιπροσωπείας αλλά και το περιεχόμενο της ε, αποστολής εκεί και της επίσκεψης. Ευχαριστώ επίσης τη Γραμματεία για το πάρα πολύ ε, πυκνό πρόγραμμα. Με τόσο καλή προετοιμασία αξιοποιήσαμε το χρόνο όσο καλύτερα μπορούσαμε. Βλέπετε ότι ήταν η αμελής αντιπροσωπεία. Αυτό δείχνει και πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Μαρτινίκα, αλλά και τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες γενικότερα. Ενδιαφέρονται πολύ τα μέλη της Επιτροπής μας για αυτές τις περιοχές και πάντα διαπιστώνουμε ότι και εκείνοι ενδιαφέρονται για τις εργασίες της δικής μας Επιτροπής. γιατί αυτές οι περιφέρειες και η Μαρτινίκα εξαρτώνται πάρα πολύ από την ευρωπαϊκή ενίσχυση ε, για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να μπορεί ο κόσμος να παραμένει, να ζει και να εργάζεται στο νησί. Επίσης έγινε και πολύ ευρεία κάλυψη στον τύπο το τοπικό και σε ό,τι αφορά τα κανάλια της τηλεόρασης, αλλά και τα, τις εφημερίδες και τα έντυπα. Ένα τελευταίο που άφησα για το τέλος, γιατί το θεώρησα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, είναι το εξή. Εκεί σταθμεύει μια μονάδα του Γαλλικού στρατού που ε, έχει δημιούργησει ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της νεολαίας. Ας πούμε, για νέους ε, που δεν έχουν ε, απολυτήριο ε, γυμνασίου έχουν κάποια προβλήματα στην κοινωνική τους συμπεριφορά και στην ένταξη, έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα από το στρατό. Ε, τους εκπαιδεύουν και, για να μάθουν διάφορα επαγγέλματα, από μηχανικός αυτοκινήτων, ας πούμε, μέχρι και, και κορίτσια επίσης, ε, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, δεν είναι μόνο για αγόρια, για να μπορούν να έχουν μια επαγγελματική κατάρτιση πάρα πολύ άρτια, επιτόπου, ε, από το στρατό και ε, από νέου ε, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς πλαισιώνονται και ως προς την κοινωνική διάσταση. Και αυτό το σύστημα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εν μέρη. Το θεώρησα πάρα πολύ καλή η δουλειά που κάνει εκεί ο στρατός και έχει και νόημα. Συμπέρασμα. Είχαμε και συναδέλφου όπως την κυρία Ροντρίγκε, που είναι από τη Μαδέρα, που είναι επίση απομακρυσμένη ε, περιοχή. Και αξιοποίησε και τις δικές της εμπειρίες και έδωσε κάποιες συμβουλές ε, και στους δόπιους. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ε, πολύτιμη αυτή η αποστολή και πολύ μας βοήθησε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας ότι συζητούμε για αυτές τις περιφέρειες, όχι μόνο στη δική μας Επιτροπή, αλλά και με άλλους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο. Έχουν μεν προβλήματα αυτές οι περιφέρειες, αλλά είναι προπομπή και φυλάκια έτσι, εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλες υπήρους και ε, προβάλλουν ε, και διαφημίζουν το κύρος ε, και το γόητρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you Ευχαριστούμε για την πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Τώρα τα μάθαμε όλα. <laughs> Η γραμματεία έχει ετοιμάσει και την έκθεση. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της αποστολής. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι το σχέδιο νομοδότησης που ετοίμασε ο εισηγητής μας, ο κ. Ζουλό, και αφορά την πρόσβαση στην χρηματοδότηση των ΜΜΕ και η αύξηση της χρηματοδότησης από, τις, από την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Η ΕΚΟΝ αποφάσισε να κάνει μια έκθεση πρωτοβουλίας ως συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου του 2013 για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση ε, σε τράπεζες και σε άλλους ε, χώρους. Ε, εμείς γνωμοδοτούμε απλώς. Ο κ. Ζουλό είναι εισηγητής της δικής μας γνωμοδότησης και σήμερα θα παρουσιάσει το σχέδιο της δικής του γνωμοδότησης. Το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΟΝ μας υποχρεώνει να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση στις 24 Μαΐου. Προτείνω ε, οι τροπολογίες να, να κατατεθούν 21 Απριλίου μέχρι το τέλος της εργάσιμης μέχρι τις 5 ας πούμε. Ο κ. Ζουλό έχει το λόγο. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάποια στοιχεία για να σας θέσω το πλαίσιο με στο οποίο κινείται η γνωμοδότηση. Όπως είπατε, αυτή η γνωμοδότηση αφορά το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως τονίσαμε ήδη στην Επιτροπή μας, στο παρελθόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και έχουν ένα δυναμικό ανάπτυξης θέσεων απασχόλησης, πολύ σημαντικό, κάποια νούμερα, για να σας δείξω ότι η ΜΜΕ σήμερα είναι 20 εκατομμύρια στην Ευρώπη και αποτελούν περίπου, ε, δίνουν 90 εκατομμύρια απασχόληση, δηλαδή το 70% το τομέα. Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης που ξεκίνησε εδώ και λίγα χρόνια, η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση ήταν όλο και πιο δύσκολη, ε, όλο και πιο περιορισμένη σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησης των ΙΜΕ από τα τραπεζικά δάνεια. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΕΚΟΝ εργάζονται επί των τραπεζικών δανείων που λαμβάνουν οι ΜΜΕ, αλλά μιλάνε και για τις άλλες πηγές χρηματοδότησης, κυρίως στα πλαίσια του σχεδίου, του σχεδίου Ένωσης Κεφαλαιογορών. Ο εισηγητής, ο κύριος Κράς, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διαφοροποίηση της χρηματοδότηση των ΜΜΕ και συμφωνώ με τη θέση του ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση της ε, πραγματικής οικονομίας και άρα και των ΜΜΕ μέσω της, ε, των κεφαλαίων αγορών. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αγορές θα υποκαταστήσουν τις τράπεζες, γιατί φυσικά οι τράπεζες συχνά ε, έχουν τις γνώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που είναι απαραίτητο για τη χρηματοδότηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, δική μου γνωμοδότηση, της Επιτροπής μας δηλαδή, στα πλαίσια του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής ΡΕτζη, επικεντρώθηκα στην εδαφική διάσταση και, και στην ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, που θα πρέπει να καταστήσουμε πολύ πιο ελκυστική. Ξέρετε ότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις είναι πάντα πολύ συνοπτικές. Άρα έχουμε δυνατότητα για να υποβάλουμε λίγες ιδέες. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας λακωνικότητας προσπάθησα να αναπτύξω την γνωμοδότησή μου παρουσιάζοντας κάποιες απλές ιδέες. Καταρχάς, διαπιστώνω ότι οι μικρομεσαίες μας κινούνται μέσα σε ένα ε, πλαίσιο που ταλανίζεται από πολυάριθμες ρυθμίσεις και κανόνες. Ε, εμείς θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο σταθερό, ξεκάθαρο, μειώνοντας ε, τους φραγμούς ε, που αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την, ε, το συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των, των διαφόρων προγραμμάτων και εργαλείων που έχουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των ΜΜΕ από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, περιφερειακή πολιτική δηλαδή, η Επιτροπή μας θα πρέπει να κάνει το παν, ούτω ώστε να προχωρήσει η απλούστευση και να δώσει και τα αποτελέσματα. Όλοι οι δικαιούχοι της πολιτικής συνοχής πλήττονται, και το είπαμε αυτό πολλές φορές, από κανόνες που είναι πολύ περίπλοκοι, υπάρχει αστάθεια, στους κανόνες αλλάζουν, ε, καθυστερούν οι πληρωμές, ε, διοικητικό άχθος, επίσης το βάρος των ελέγχων είναι πολύ επαχθές και οι επιχειρήσεις γενικά, αλλά και οι ΜΜΕ, ε, κυρίως πλήττονται ακόμα πιο σκληρά, γιατί κινούνται μέσα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο και η ανάγκη να δοθούν αυτά τα κονδύλια ε, δημιουργούν πολλά προβλήματα στα ταμεία τους. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ρευστότητα στα ταμεία. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις πολλές από αυτές τουλάχιστον δεν έχουν τις απαραίτητες ε, υπηρεσίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά το κόστος διαχείρισης είναι δυσανάλογο συχνά σε σχέση με τα ποσά για τα οποία μιλάμε. Και ακριβώς γι' αυτό πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προτιμούν να στραφούν απευθείας στις τράπεζες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται από τις αντιφάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην περιφερειακή πολιτική και στην πολιτική ανταγωνισμού από την άλλη και ακριβώς γι' αυτό στην έκθεσή μου ζητάω από την Κομισιόν να διευκρινίσει την σχέση που υπάρχει μεταξύ της πολιτικής συνοχής από τη μία και των κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις από την άλλη. Τέλος, τελευταίο σημείο. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που καθορίζουν τη φύση και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε ΜΜΕ στο, στο τέλος της αλυσίδας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν πολύ, πολυπίκυλες παραμέτρους. Η δική μας Επιτροπή μπορεί να παίξει μια, ένα ρόλο και να εξασφαλίσει μια προστιθέμενη αξία για να κρατήσουμε υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες των ΙΜΕ, τόσο ώστε να προσφέρει ε, δεδειγμένες λύσεις χρηματοδότησης. Ένα βασικό στοιχείο είναι το μέγεθος της ίδιας επιχείρησης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες λοιπόν των επιχειρήσεων ας πούμε. Αλλά δεν είναι το μόνο θέμα αυτό, η μόνη παράμετρος. Φυσικά, ο χώρος, το πλαίσιο, το που βρίσκονται οι μικρές επιχειρήσεις έχει μεγάλη σημασία. Οι συνθήκες ε, η χρηματοδότηση, α πούμε, στη Γουαδελούπη ή στη Μαρτινίκα, φυσικά δεν είναι το ίδιο με αυτέ στο Παρίσι. Και φυσικά, πέρα από το μέγεθος, πέρα από την ε, περιοχή, υπάρχει και ο τομέα ε, δραστηριότητας, το επιχειρηματικό μοντέλο, η νομική μορφή που έχουν αυτέ οι επιχειρήσει μεταξύ αυτών των παραμέτρων υπάρχει και η φάση κύκλου. Σε τι φάση είναι η επιχείρηση, στη φάση της ανάπτυξή της δηλαδή. Θα πρέπει η περιφερειακή πολιτική να είναι σε θέση να δώσει λύσεις ενδεδειγμένες, κατάλληλες, όχι μόνο για να δημιουργηθούν ας πούμε οι επιχειρήσεις, όχι μόνο για να υπάρξουν οι start-up, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά για να μπορέσουν και να επιβιώσουν συνεχεία και να μεγαλώσουν. Και για να σας αποδείξω αυτά που λέω, σε ορισμένε περιπτώσεις τα χρηματοδοτικά εργαλεία ε, είναι κατάλληλο μέσο, αλλά μερικές φορές οι παραδοσιακές επιδοτήσεις είναι καταλληλότερες, ανάλογα με τις ε, συνθήκες. Καταληκτικά. Δεν έχουμε δυστυχώς σε μια τόσο σύντομη γνωμοδότηση να βάλουμε όλες τις ιδέες που υπάρχουν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο μπορεί και εγώ ο ίδιος να τροποποιήσω τα, το κείμενό μου και φυσικά θα ακούσω και όλες τις παρατηρήσεις από τους συναδέλφους για να εμπλουτίσω περαιτέρω την γνωμοδότηση και να λάβω υπόψη τις προτάσεις τους. Είτε τώρα είτε αργότερα, όταν κατατεθούν οι τροπολογίες δηλαδή. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε την συζήτηση και με τους σκιώδεις εισηγητές. Ο κ. Πίκολα καταρχήν. Ο κ. Πίτσουλα λοιπόν. Ευχαριστώ τον κύριο Ζουλό για το προσχέδιό του περί πρόσβαση ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την αύξηση της πολυμορφίας χρηματοδότηση. Συμφωνώ ότι οι μικρομεσαίε επιχείρησει ε, είναι η ατμομηχανή στην δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζω την, ε, το γεγονό ότι η πολιτική συνοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περίοδους περικοπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αποτελούν το 90% των ε, επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γεννούν τα 2 τρίτα των θέσεων εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αντιπροσωπεύουν πάνω το 50% της προσθέμενης αξίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 άτομα προσωπικό. Συμφωνώ με την εκτίμηση ότι οι μικρομεσαίε επιχείρησει θα πρέπει να έχουν πιο ε, εύκολη πρόσβαση στα κεφάλαια. Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαθεσιμότητα κεφαλαίων και επιστώσεων είναι το σημαντικότερο μάλιστα πρόβλημα των επιχειρήσεων που δεν βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να τονίσει την σημασία να διαθέτουν χρηματοδότηση ιδιαίτερα σε περιοχές όπως νησιωτικές ε, ή ορεινές περιοχές. Εκεί η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται επίσης και από υψηλό διοικητικό άχθος, εκτός της δυσκολίας στην πρόσβαση. Άλλο πρόβλημα είναι ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός τέτοιων επιχειρήσεων ε, δρούν ε, διασυνοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους και πρόσθετες δυσκολίες ε, που τις εμποδίζουν στο να υλοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν το δυναμικό τους. Γι' αυτό το λόγο και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα και να καταστήσουν πιο ελκυστική την επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την έκθεσή του και θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Πρόεδρος, δεν βλέπω σκιό εισηγητή από το ECR και τους φιλελεύθερους. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν είναι εδώ εισηγητής μας, μιλώ εκ μέρου του. Μας, ε, αρέσει, μας αρέσουν ιδιαίτερα δύο πράγματα, δύο σχόλια για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ε, πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε ιδιαίτερα εμεί στην ECR, και δεύτερον, ότι δεν θα πρέπει να κατασταθεί ο ρόλος των τραπεζών. Ε, αυτή η, η, διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται, η πολυμορφία θα πρέπει να είναι πρόσθετη έναντι των, του ρόλου των τραπεζών. Θα έχουμε και άλλα σχόλια στο μέλλον. Ευχαριστώ. της κυρίας Νικολάη, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα. Να πω τα εξή. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αποθαρρύνονται από το διοικητικό άκθος που συνδέεται με την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Οπότε θα πρέπει η πρόσβαση στη χρηματοδότηση να γίνει με μεγαλύτερη διαφάνεια και με πιο απλό τρόπο. Η κυρία Νικολάη λοιπόν ε, συμφωνεί με τον ορισμό της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου ε, για τη μείωση της γραφειοκρατίας ε, στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διαστατικών Ταμείων και περιμένουμε τις ε, ε, συστάσεις της. Δεύτερον, το δίκτυο επιχείρηση στην Ευρώπη, επιχειρήση στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και για το πώς αυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, τις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης που τους παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εθνικό επίπεδο αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να γίνονται, να κοινοποιούνται και να είναι διαθέσιμες. Οπότε και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μονοπευθυντικές θηρίδες όπως το δίκτυο Enterprise in Europe. Τρίτο σημείο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, εναλλακτική πρόσβαση χρηματοδότηση με πιο απλό τρόπο. Ε, η Ένωση, Κεφαλαίου η Ένωση Κεφαλαιογορών είναι ένα σημαντικό εργαλείο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ισότητα ευκαιριών σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις επιχειρήσεις. Οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ διαφορετικές και επικοινόμορφε. Δεν υπάρχει μία βέλτιστη πρακτική. Η κυρία Νικολάη συνεπώς βλέπει, ότι εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και με καινοτόμο τρόπο ε, τις ε, σύγχρονες ε, τεχνικές χρηματοδότησης όπως τη FinTech διότι ε, μέσω αυτής μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν ενδεχόμενους εταίρους. Θα υποβάλει και τροπολογία για αυτό το θέμα. Τέλος, η κυρία Νικολάη ορίζει την ε, έκκληση του εισηγητή της ΕΚΟΝ προκειμένου τα ε, κράτη-μέλη να βελτιώσουν την οικονομική επιμόρφωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπογραμμίζει επίσης ε, το ότι μια εξειδικευμένη εκπαίδευση θα μπορούσε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Βάνα, εξ ονόματος της ναι, ζητώ συγγνώμη Ντάβος Κάρα από την ομάδα των Πρασίνων δυστυχώς κολλείται. Θέλει να πει ότι χαίρεται για την άφορα που γίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή εκτός από αναφορά στο γενικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζουλό για την εξαιρετική του γνωμοδότηση. Συμφωνούμε ότι ο συντονισμός, η συνέπεια και η συνέργεια μεταξύ των προγραμμάτων και των ε, μέσων που υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι δεδομένα. Θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία που έχουν ε, οι μικρομεσαίες για την ευρωπαϊκή οικονομία και πόσο μπορούν να αυξήσουν και να τονώσουν την ανάπτυξη και την μεγέθυνση. Θα πρέπει εδώ να ενταχθεί και η αρχή της κυκλικής οικονομίας για να φτάσουμε σε αυτό το σκοπό και να δημιουργηθούν λεγόμενες πράσινες θέσεις εργασίας. Είναι πολλές οι ευκαιρίες για καινοτομία και μπορούν να μεταφραστούν σε μόνιμες και καλές δουλειές ε, με πράσινους διαγωνισμούς για τα δημόσια έργα, έτσι θα στραφούν και θα προσανατολιστούν προς τη σωστή κατεύθυνση μικρομεσαίες. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι και η ευφορία και η βιωσιμότητα των τοπικών αγορών και πώς μπορούν και να συνεισφέρουν τα ευρωπαϊκά διαρθωτικά και επενδυτικά κονδύλια. Θα ήθελα επίσης επ' να θυμίσω και πάλι ε, το πρόβλημα που έχουμε ε, με το φύλλο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ας πούμε και στην αντίστοιχη πράξη. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν ε, μεγαλύτερη προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτό το σημείο μέχρι να αρχίσουμε να βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Thank you, thank you very much. The next shadow, ευχαριστώ. Η κυρία Νταμάτο, επόμενη σκιώδη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η έκθεση του κυρίου Ζουλό είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εμείς στην Επιτροπή ΡΕΤΖΙ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς αναπτύσσονται οι ΜΜΕ και εμένα κυρίως ως εισηγήτρια μια έκθεση για τον θεματικό στόχο 3 και επομένω την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Ο συνάδελφος τονίζει ότι οι ΜΜΕ έχουν πρόβλημα ε, με την περιπλοκότητα της νομοθεσίας και το διοικητικό άχθος ε, για την πρόσβασή τους ε, στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Ζητούμε λοιπόν μια βαθιά πλούστευση από την Κομισιόν και να διευκρίνει τη σχέση ανάμεσα στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και στις κρατικές ενισχύσεις. Συμφωνώ επίσης και με την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τη συνέργεια, το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα διάφορα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγώ το κήρυμα Cinque Stelle έχουμε διάφορα προβλήματα για την πρωτοβουλία της Ένωσης Κεφαλαγορών. Είναι ένα σύνολο πρωτοβουλειών που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν το σκιώδες λεγόμενο τραπεζικό σύστημα και άρα τα μη τραπεζικά δάνεια. Ε, θα πρέπει να δούμε τις υποδομές ε, κυρίως και τις, της Ένωσης Κεφαλαγορών και το πόσο καταλάλληλες είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιογορών, αν είναι αναρμονισμένοι, οι δυνατότητες να έχουν πρόσβαση οι πολίτες και οι ΜΕ σε χρηματοδότηση, η δυνατότητά τους διευρύνεται. Φυσικά αυτό εξαρτάται από το κράτος μέλος, δεν εξαρτάται, δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το κράτος μέλος το οποίο ε, διαμένουν. Ε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι μακροπρόθεσμα τι όφελος θα έχουν οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, μία από τις προτεραιότητες της Κομισιόν είναι η εξή. Η πρατική ε, παραχώρηση ενός χαρτοφυλακίου που έχει παραχωρήσει μία τράπεζα και συνεχεία μπαίνει στην αγορά. Ε, και συνεχεία μπαίνουν, ε, γίνεται αυτό, αυτό το χαρτοφυλάκιο ας πούμε, τίτλοι ε, τιτλοποιείται α πούμε και μπορεί να πουληθεί σε επενδυτέ. Αυτό όμω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κατά τη γνώμη μα. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οι επενδυτέ αγοράζουν αυτού του τίτλου και πληρώνονται μόνο εάν τα δάνεια τα οποία εμπεριέχονται στους τίτλους αυτού πληρωθούν. Αυτή η τεχνική ήταν η ουσία της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Από εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή οι τράπεζες μπορούσαν ε, τα τοξικά δάνεια ε, κακής ποιότητας ας πούμε, να τα τιτλοποιήσουν ε, και ε, συνεχεία να πάρουν και το rating, ας πούμε, αλφα-αλφα-αλφα ή πολύ καλή βαθμολογία, Η Κομισιόν θα πρέπει να μας εξηγήσει ποια είναι η καλή τιτλοποίηση μέσω μια σειράς από κριτήρια που, καθιστούν την τιτλοποίηση πιο απλή και πιο διαφανή. Η δημιουργία όμως νέων τίτλων, ε, η παροχή εγγυήσεων και όλα αυτά παρέχονται από τις επενδυτικές τράπεζες, το να ιδιωτικοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία, αυτό προωθεί στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα των επενδυτικών τραπεζών σε σχέση με την παραδοσιακή ας τραπεζική σχέση που, που, που ξέραμε. Μην ξεχνάμε εδώ το ρόλο που είχαν ε, οι επενδυτικέ τράπεζε στη χρηματοπιστωτική κρίση. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει η παραδοσιακή τραπεζική σχέση να διατηρηθεί ω ο βασικό τρόπο ε, εξασφάλιση πίστοση από τι ΜΜΕ. Και αυτό θα πρέπει να προτιμάμε κανεί. Θα πρέπει να προτιμάμε η ΜΜΕ. Ε, ο συνάδελφο είπε ότι τα τραπεζικά δάνεια χρειάζονται ε, για να βελτιωθεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και για να κάνουν ε, πιο ενδιαφέρουσες τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσει για τις ΜΜΕ. Αλλά το να μεταφέρουμε τις, τους κινδύνους από τις τράπεζες σε ιδιωτικούς ας το σύστημα δεν γίνεται πιο ασφαλές και μπορεί να δημιουργηθούν νέα επίπεδα ας πούμε, ηθικού κινδύνου. Και κάποια στιγμή θα χρειαστεί πάλι να ξανασώσουμε ας πούμε, τις τράπεζες ε, με τα λεφτά του φορολογούμενου. Το βασικό θέμα είναι ε, μέσω της χρηματοδότησης ε, να εξασφαλίσουμε μείωση της ε, ανεργίας, να εξασφαλίσουμε το διαχωρισμό ανάμεσα στην επενδυτική τράπεζα και στην παραδοσιακή τράπεζα, ούτως ώστε να είναι πιο ανθεκτικά γενικά οι τράπεζες. Ευχαριστώ. Ακολουθούν οι υπόλοιποι Ο eh, Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις πιστώσεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε προσεκτικά το πώς είναι δυνατόν να διευκολύνουμε την ε, ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η τράπεζε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, έχουμε δει συγχωνεύσεις τραπεζών, οι οποίες δημιουργούν ε, τεράστια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ε, με ε, οι οποίες ε, όμως εστιάζουν στις μεγάλες πόλεις ενώ στις αγροτικές και στις εξωαστικές περιοχές δεν υπάρχει ούτε ένα υποκατάστημα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση οι μικρόμεσες επιχειρήσεις εκεί. Θα πρέπει να βρούμε καινούρια, τρόπο, καινούρια μέσα λοιπόν όπως η... Ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών ε, για να καλύψουμε το κενό αυτό των τραπεζών. Είναι μια συζήτηση η οποία θα πάρει χρόνο όμως. Μετά, ε, η νομική μορφή. Σε ορισμένες χώρες μιλούμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σαν να είναι ένα ενίο πράγμα. Στην πραγματικότητα Υπάρχουν πολλοί τύποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχουν και διαφορετικές ανάγκες χρηματοδότησης. Το 10% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη δεν είναι ανώνυμες εταιρείε. Ε, είναι συνεταιρισμοί, οι συνεταιριστικές εταιρείε που Εξαιτία τη νομικής του ε, φύση, ε, τη νομική μορφής, δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένε μορφές, χρηματοδότηση. Όμω, το ευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλε τι μικρομεσαίε επιχείρησει ανεξαρτήτω νομικής μορφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρέσο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Ζουλό είπε πάρα πολλά πράγματα. Διερωτώ αν μιλήσετε για το δυναμικό που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να εκμεταλλευτούν το σχέδιο Juncker. Ένας από τους βασικούς άξονες του σχέδιου Juncker ήταν ακριβώς οι ίδιες οι μικρομεσαίες. Έχετε κάποιες ε, ειδήσει για το τι συμβαίνει με τον άξονα αυτό του σχεδίου Juncker. γιατί θα, και μπορούσε και αυτή η Ένωση Κεφαλαιογορών να χρησιμοποιηθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μέσω της ε, έτσι, διερεύνησης νέων εργαλείων. Διερωτώ με, τι απέγινε αυτό το σημείο. Επειδή δεν έχετε πολύ χώρο στην εκθεσία σας δεν το αναφέρετε. Τέλο εσείς το έχετε ψάξει καθόλου. Έχετε ειδήσει, πληροφορίες. Επόμενο you, Mr. ο κύριος Νοβάκοφ. Thank you very much, First of all, uh, I'd like to... Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ζουλό για τις ε, προσπάθειές του. Η έκθεση του είναι ισορροπημένη. Θα ήθελα να ε, στηρίξω τη γνώμη του, τη αυτή και ιδιαίτερα να τονίσω την ανάγκη απλοποίησης και μείωση της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που διάβασα, το 70% των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πιστέψουμε τους 7 στους 10. Είναι μια σημαντική πλειοψηφία Ορισμένοι προηγούμενοι ομιλητέ ε, είπαν ότι υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης, έλλειψη πόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι αλήθεια αυτό ακριβώς. Υπάρχει ε, έλλειμμα πρόσβασης, όχι έλλειμμα κονδυλίων. Το προγράμματα του προγράμματος και σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο ε, υπάρχουν αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν ε, αίτηση να υποβάλουν πολύ περισσότερο να διαχειριστούν τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα. Γνωρίζω ε, αρκετά παραδείγματα σε περισσότερες από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν ε, συγκεκριμένα εργαλεία για νότευκτες επιχειρήσεις. Ακόμα και για αυτές όμως υπάρχουν ε, υποχρεώσεις. Ε, αν αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν την οικονομική και διοικητική ικανότητα, δεν μπορούν καν να υποφεληθούν των εργαλείων αυτών. Ε, αυτό όμως είναι δύσκολο σε νέες επιχειρήσεις, σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα λοιπόν. Ε, επίσης θα πρέπει να επι Ταχύνουμε τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε άλλο αυτό. Επισήμως το κόστος διαχείρισης των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ανέρχεται στο 8% του προπολογισμού του προγράμματος. Πιστεύω ότι στην πράξη είναι περισσότερο αν λάβουμε υπόψη τους συμβούλους, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ ίσως ξεπερνάει και το 10%. Φαντάζεστε να έχετε ένα σύστημα άρδευσης που ε, σπαταλά ένα στα 10 λίτρα. Αναποτελεσματικότατο. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι να κάνουμε έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσει τα πορίσματά της πριν μάλιστα το ε, τέλος των εργασιών της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Νόβακοφ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι καλό σημείο αφετηρία η έκθεσή του, η γνωμοδότησή του. Να δούμε πόσο μπορούμε και πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Να σας επιστήσω την προσοχή σε δύο πτυχές του θέματος αυτού στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους τομείς όπου το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί. Δεν ε, βοηθάει δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εκεί ακριβώς θα μπορούσαμε να δώσουμε εναλλακτικέ λύσει Μέσω διαφόρων εργαλείων. Δάνεια, εγγύησει κτλ. Αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε διάφορα μέρη στην Ευρώπη. Γιατί όταν οι τράπεζε βλέπουν ότι υπάρχει ανταγω... Ε, κάποιος στο δημόσιο τομέα με τη χρήση των διαφθορτικών ταμείων, τότε μειώνουν και τις προσδοκίες ε, να βγάλουν κέρδος ε, από τα δάνεια που δίνουν, δηλαδή μέσω μεγάλων επιτοκίων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικά χρειάζονται γρήγορη ε, και φθηνή χρηματοδότηση, ώστε να μεγενθηθούν, να αναπτυχθούν. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση επίσης και στην απλούστευση των διαδικασιών όταν ε, προσπαθούν οι επιχειρήσει να βρουν λεφτά από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ο χρόνος διεκπαιρέωση των αιτήσεων αυτών θα πρέπει να μειωθεί. Συχνά οι επιχειρηματίες, καθώς περιμένουν και του έρχεται απάντηση, τελικά παρετούνται από αυτή την προσπάθεια, α πούμε, γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος να πάρει κανεί λεφτά από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Και απλώς παρετούνται από αυτό το μέσον. Μερικέ φορές οι εταιρείε πρέπει να δράσουν πάρα πολύ γρήγορα. Εάν χρειαζόμαστε μια αιωνιότητα για να βρούμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποιο θα ασχολείται. Αν υπάρξει απλούστευση, παραδείγματο χάρη τα κονδύλια από το, τον ορίζοντα 2020 και το κόσμο, αν δούμε πόσε εταιρείε παίρνουν λεφτά από αυτά τα προγράμματα και πώ, βλέπουμε ότι μόνο ελάχιστες μικρές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα τελικά. Γιατί όλη η διαδικασία είναι πάρα πολύ επαχθής για να πάρει κάτι λεφτά έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανίς Ρόη. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μόνο τρία πράγματα συμπληρωματικά. Ίσως να ήταν φρόνιμο στο σημείο 5 να, πούμε το εξή εκεί λέει ότι υπάρχουν διαφορές ανάλογα με την ανάπτυξή σου, τον κλάδο σου και την έδρα σου. Οι διαφορές στην έδρα και στις περιφέρειες ε, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι να υπάρχει μία έκθεση υλοποίησης ή εφαρμογής για να δούμε ποιος αντλεί διάφορα κονδύλια και ποιος τα απορροφά σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ε, γίνεται λόγος ε, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια ένωση κεφαλαίου αγορών. Αυτό είναι συνολικό, είναι καθολικό σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως τεράστιες διαφορές. Αν είσαι σε μια χώρα που έχει ακόμα πολλά προβλήματα μετά από τη χρηματοοικονομική κρίση, είναι πολύ πιο δύσκολο να έχεις πρόσβαση σε κονδύλια ε, σε σύγκριση με κάποιον που βρίσκεται στις κάτω χώρες, για παράδειγμα. Θα μπορούσε κάποιος να μας κάνει μια έκθεση, τι γίνεται με τις διάφορες ε, χώρες στην Ευρώπη, με τις διάφορες περιφέρειες, αναχώρα ή αναχώρα ε, σύγκλησης, περιφέρεια σύγκλησης, για να έχουμε μια στοιχειώδη ιδέα. Αλλιώς παραμένει πάρα πολύ γενικόλογο αυτό. Και δεν προχωρούμε. Αυτό που λέει το σημείο 5, ας πούμε, έχετε δίκιο να το λέτε έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ ακόμα ασαφές και γενικό. Ε, για να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτό και μετά ε, πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ε, τα διάφορα εργαλεία μας. Η ΕΚΟΝ νομίζω κινείται σε πάρα πολύ γενικά πλαίσια και ασαφή και αόριστα. Εμείς θα πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο. Στη συνέχεια, στο σημείο 4 μιλάτε για τις κρατικές ενισχύσεις. Ωραία. από τον ορίζοντα 2020 ας πούμε υπάρχει στήριξη χωρίς κανένα πρόβλημα για τις εταιρείε, τα προβλήματα όμως παραμένουν αλλού με τους ελέγχους. Εσείς μιλάτε για διευκρινήσεις, για εξακρίβωση που υπάρχουν τα προβλήματα για να τα λύσουμε. Συμφωνώ 100% μαζί σας να αναφερθεί και αυτό. Και ένα τρίτο και τελευταίο Διστάζω ακόμα με τον ορισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ποιοι, τι είστε η μικρομεσαία επιχείρηση, τι είναι νεοφυής, ε, τι είναι επιχείρηση που ζητάει χρηματοδότηση και έχει λιγότερους από 10 εργαζομένους. Ε, λοιπόν, αν είσαι μια επιχείρηση που τώρα ε, ακόμα προσπαθείς να σταθείς στα πόδια σου και δεν έχεις 10 εργαζομένους, δεν σημαίνει ότι είσαι μικρομεσαία. Αν είσαι, ξέρω εγώ, μια εταιρεία που έχει 4 με 8 εργαζομένους, είσαι μια πολύ μικρή επιχείρηση που έχεις δυσκολίες χρηματοδότησης και δεν εμπίπτεις και γενικότερα σε ένα ορισμό. Θα κάνω και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή για να διευκρινίσουμε κάπως τα πράγματα στη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, thank you very much. And the last question... Ο κύριος Πότσακ, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω από αυτό που είπε ο συνάδελφος Νοβάκοφ και ο συνάδελφος Χέτμαν. Και αυτό έχει να κάνει με ε, το γραφειοκρατικό άχθος. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να έχουμε σταθερότητα, ένα συγκεκριμένο σταθερό νομικό πλαίσιο ε, που να μπορεί κανείς να ε, επαφίεται σε αυτό να υπάρχει σταθερότητα και αξιοπιστία με λίγη γραφειοκρατία και ε, με απλές διαδικασίες που να μην αλλάζουν συνέχεια. Και σε σχέση με όλα αυτά πιστεύω ότι για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σταθερό νομικό πλαίσιο ε, είναι απαραίτητο να ε, επέλθει αυτή η απλούστευση που ζητάμε κι εμείς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, ε, ή θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με μέλη της ομάδας υψηλού επίπεδου και να τα τονίσουμε ξανά αυτά τα θέματα. Παρόλο που ξέρω ότι υπάρχουν και περιορισμοί χώρου και μήκου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουλό, εισηγητής, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει. Oui, ασφαλώς, ευχαριστώ. Θα πω δύο λόγια αλλά σύντομα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω του κοιόδης ηγητές που πήραν το λόγο, αλλά και τους συναδέλφους, υπόλοιπους συναδέλφους, για τι προτάσει του, για τι ε, παρατήρησει του. Όλα αυτά δείχνουν το ενδιαφέρον μας ε, ως Επιτροπής για την ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θα σχολιάσω όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Τι σημείωσα. Σημείωσα αυτά που αποσχολούν τον καθένα σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση σε κεφάλαια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το διαφορετικό χαρακτήρα μεταξύ των διαφόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετέχει το θέμα του ορισμού, δεν υπάρχει ορισμός του τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια διαφέρουν και ανάλογα με το πού είναι εγκατεστημένες. Ένα άλλο θέμα το οποίο υπογραμμίστηκε επανειλημμένως είναι η απλοποίηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρόσκομα. Τρίτον, η συμπληρωματικότητα μεταξύ χρηματοδότηση από τράπεζες και χρηματοδότηση από τις ε, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη αυτής της ποικιλομορφία, ε, ε, συμπληρωματικότητα με διαφάνεια μεταξύ αυτών των μορφών χρηματοδότησης. Πέμπτον, η ασφάλεια των προϊόντων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στην, στις κεφαλαίες αγορές με ασφαλή τρόπο. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο Juncker, πάνω από 20 σχέδια ε, υπογράφηκαν από βράση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Γαλλία τουλάχιστον ε, περιλαμβάνουν 30.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ βέβαια ε, θα γνωμοδοτήσει επί της οπότε εγώ δεν το ανέφερα διότι θεωρώ ότι βρίσκεται στη δική τους αρμοδιότητα. Αλλά πάντως ε, στο κομμάτι αυτό ήταν χρήσιμες οι παρατηρήσεις σας. Ε, περιμένω και τις τροπολογίες σας και τις συγκεκριμένες προτάσεις σε κείμενο έτσι ώστε να τις συμπεριλάβω στην ε, δική μας γνωμοδότηση. Πρόεδρος, κατά δεν έδωσα το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη θα έπρεπε να το είχα κάνει πιο νωρίς. Θα το κάνω τώρα όμως. Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο. Καταρχήν, ποιος θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Αλέξη Μαρσόν από τη Γενική Διεύθυνση Φίσμα. Δύο λόγια για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και το πρόγραμμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε ένα πρόγραμμα δράσης για τη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών το Σεπτέμβριο του 2015. Μία από τις βασικές προτεραιότητες αυτού του πρόγραμματος δράσης είναι ακριβώς η διευκόλυνση της ε, ε, πρόσβασης στη χρηματοδότηση από πλευράς επιχειρήσεων και ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος είναι να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση από πλευρά τραπεζών με ένα και δεύτερο σύστημα ε, που θα δίνει ε, διάφορε, διάφορες ε, δυνατότητες όπως για παράδειγμα για τις νοφίες επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα δράσης συμπεριλαμβάνει μια σειρά δράσεων για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Να σας πω τρία, σας δώσω τρία παραδείγματα τέτοιων δράσεων. Πρώτον, ένα πακέτο για να προωθήσουμε τα κεφάλαια ε, κινδύνου. Για παράδειγμα με τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ε, ταμείου ταμείων για το που θα παρέχει δηλαδή κεφάλαια κίνησης θα αποτελέσει δηλαδή ένα ειδικό όχημα για τέτοιου είδους κεφάλαια. Δεύτερον, ε, δράσεις για την καλύτερη ε, σύνδεση επιχειρήσεων που θα έχουν ε, πιο μεγάλες δυνατότητες χρησιμοποίησης των χρηματοδότησης, δηλαδή θα τους δώσουμε τη δυνατότητα σε εναλλακτική χρηματοδότηση, ε, λαμβάνω υπόψη την ιδέα της δημιουργίας μονοπευθυντικών θηρίδων ε, σε εθνικό επίπεδο, που θα δίνουν προφορίες για τέτοιου είδους πηγές χρηματοδότησης. Τρίτον, τη αναθεώρηση της οδηγίας εγχειριδίων. Ένας από τους στόχους θα είναι οι απαιτήσει να είναι λιγότερες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις, μικρομε... για τις μεγαλύτερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουλάχιστον, ε, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε λίγο τις αγορές και, ε, ε, και τις κεφαλαίες σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η, DG, η Γενική Ρίτζιο δεν θέλει το λόγο. Ωραία. Ευχαριστώ. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω ότι προτείνουμε ε, ε, οι τροπολογίες να έχουν κατευθεί μέχρι τις 5 το απόγευμα, 5η 21 Απριλίου. Αυτή είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ε, σχέδιο γνωμοδότησης της ε, Κωνσταντς Κρέλ, προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του πολιετούς μεσονομικού πλαισίου 2014-2020, η συμβολή του Κοινοβουλίου εν ώψη της πρότασης της Επιτροπής. Ο κανονισμός για το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο αναφέρει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια ε, αναθεώρηση της λειτουργίας του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου μέχρι το τέλος του 2016 το αργότερο. Η Επιτροπή Προπολογισμών αποφάσισε ε, να ε, εκπονήσει μια στρατηγική γνωμοδότηση πρωτοβουλία προκειμένου η Επιτροπή να γνωρίζει εκ των προτέρων τα θέματα για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε ε, να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση. Η Επιτροπή μας προετοιμάζει μια γνωμοδότηση. Ε, η κυρία Κρέλ είναι η συγγήτριά μας και θα μας ε, παρουσιάσει το προσχέδιο γνωμοδότησης της. Μεταξύ άλλων θα καλύπτεται από την αναθεώρηση η η αποτελεσματικότητα των, της δωρεάν ενίσχυσης σε σχέση με άλλους μορφές χρηματοδότησης, τα προκατανεμημένα εθνικά κονδύλια, ε, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός επταετούς προγράμματος κλπ. Ε, είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση έτσι ώστε ε, να ψηφίσουμε τη γνωμοδότησή μας και πάλι στις 24 Μαΐου, στις 24 Μαΐου λέω, οπότε η προθεσμία τροπολογιών είναι και πάλι 21 Απριλίου. Ε, θα έχουμε χρόνο όμως ανταλλαγής απόψεων σήμερα. Κυρία Κρέλα, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για μένα η αρχή της εβδομάδας είναι, πώς να το πω, λίγο περίεργη γιατί για πρώτη φορά προσγειώθηκα και πάλι πριν από δύο ώρες στο αεροδρόμιο των Βρυξελών όπου πραγματικά δεν επικρατεί η κανονικότητα. Είναι λίγα και τα αεροπλάνα και λίγος ο κόσμος και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εξίσου και έχει σημασία στο Κοινοβούλιο να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας κανονικά για να έχουμε μια αίσθηση κανονικότητας και να δείξουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι από τη μια μπορεί να είναι κάτι τρομακτικό ή τρομοκρατικές ε, επιθέσεις, αλλά δεν επηρεάζουν τη δουλειά μας. Αλλά δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όπως κανείς ε, φαντάζεται. Ας έχει όμως, όπως και να έχουν τα πράγματα, θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου για την ε, μεσοπρόθεσμη ε, υπόθεση αυτή του Πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, το είπατε και εσείς Πρόεδρε, θέλω να πω το εξή στη συζήτηση για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, παίζει ρόλο και ε, ε, το θέμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα και άρρηκτα συνδεδεμένα. Και στην γνωμοδότησή μου θα βρείτε μερικά σημεία όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι κανονικά αυτό ανήκει στην ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής. Αλλά επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη συνάφεια, τα δύο είναι πάγια τακτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων να τα συνδέει και να υπερασπίζεται την πολιτική συνοχή απέναντι σε διαφόρους που θεωρούν ότι α, είναι υπερβολικός ο υπολογισμός και έχουμε πολλά λεφτά εμείς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά πολύ καλύτερα αλλού αντί για την πολιτική συνοχή. Γι' αυτό στην γνωμοδότησή μου θα βρείτε και τα δύο να τα αναφέρω και να τα υπερασπίζομαι. Δεύτερον, να κάνω μια παρατήρηση Μακάρι να είχα διπλάσιο και τριπλάσιο ε, χώρο για τη γνωμοδότηση αυτή. Δηλαδή, ορισμένα θέματα τα αναφέρω μόνο επιγραμματικά, γιατί δεν χωρούσαν. Θα κάνω και τροπολογίες ε, προσωπικά για να τα συμπληρώσω. Και δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω τους συναδέλφους να το πράξουν και εκείνοι. Διότι σε μια σελίδα τι να πρωτοπείς. Ε, δεν χωράει τίποτα παραπάνω από όσα ήδη έχει γραμμένα η σελίδα ξέρω ότι υπάρχουν σημεία που μπορούμε να εμπαθύνουμε. Όπως βλέπετε, αρχίζω τη γνωμοδότησή μου και πάλι ε, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι αυτός σκοπός. Το θέμα δεν είναι να, κόβουμε κορδέλες για να κάνουμε ωραία εγγένεια ωραίων έργων που έχουν ολοκληρωθεί, ε, υποδομών και άλλων, αλλά είναι ε, ένα πρόγραμμα επενδυτικό για την περιφέρεια, για να τους δώσουν πνοή ε, των περιφερειών, ανεξαρτήτως κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Έχουμε περιφέρειες που χρειάζονται μεγάλη ενίσχυση, υπάρχουν και άλλες περιφέρειες που πηγαίνουν πολύ καλά οικονομικά και παρόλα αυτά χρειάζονται ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένα έργα πάντα. Και η πολιτική συνοχή είναι και παραμένει το μοναδικό μέσο και εργαλείο που ερμηνεύει τη συνοχή, τη συνάφεια και την αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών και την εφαρμόζει στην πράξη ενεργητικά. Γι' αυτό στην γνωμοδότησή μου υποστηρίζω θερμά το εξή. Παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τη νέα προγραμματική περίοδο, ε, τονίζω ότι δεν θα πρέπει να μειωθεί ο προπολογισμό τη πολιτική συνοχή. Δεν το επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Στη δική μου γνωμοδότηση επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι σημαντικό βήμα ήταν ε, το γεγονό τη συγχώνευση των πέντε ταμείων όχι μόνο το περιφερειακό, το συνοχής και το κοινωνικό, αλλά και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΦΕΝΤΕΡ και το Ταμείο Αλίας. Είναι καλό που όλα αυτά μπήκαν σε έναν κορβάνα και χαίρομαι που τους τελευταίους μήνες διάφορα έργα ε, που ανήκουν εδώ τα έχω επισκεφτεί προσωπικά και πραγματικά αποδίδει και πιάνει τόπο αυτή η συγχώνευση και πραγματικά δημιουργείται και συνέργεια και βελτιώσεις έχουμε από τη συνένωση των ταμείων. Καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, πώς χρηματοδοτούνται. Τώρα δεν είμαι βέβαια αν αυτό έχει γίνει παντού, αλλά είναι θετικά, πάρα πολύ θετικά τα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Και καλό είναι να το λέμε γιατί το θέμα της αποτελεσματικότητας των πόρων τον πιάνουν τόπο εάν είναι στραμμένα προς συγκεκριμένα αποτελέσματα θα μας ε, συνοδεύει και στο μέλλον Μα συνοδεύει και από την αρχή της περίοδου και δεν είναι θέμα μόνο ότι αυτό το θέτουν ελεγκτικά όργανα. Θέλουμε και εμείς να βλέπουμε αποτελέσματα, να προχωρούν οι περιφέρειες και όχι να γίνονται έργα για τα έργα και να πιάνουν τόπο και να απορροφούνται όλα τα κονδύλια. Και στη γνωμοδότηση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε απλοποιημένη πρόσβαση στα κονδύλια. Να το ξανατονίσουμε αυτό, γιατί στο μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον, πώς το λέτε, έχει συστήσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου που κάνει τις πρώτες ε, προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές. και μερικές από τις ιδέες που είχαμε ε, βάλει εμείς στο γενικό κανονισμό αποδίδουν με τα καταποκοπή ποσά που επιτρέπουμε και στο Κοινωνικό Ταμείο και στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ήδη αποδίδουν κάποιους καρπούς, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά περισσότερα έτσι ώστε να βελτιωθεί και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των κονδυλίων. Και όπως ακούσαμε και προηγουμένως από την πρώτη έκθεση, στην πρόσβαση για τις μικρομεσαίες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να το ξαναπούμε και να το ξεκαθαρίσουμε ότι χρειάζεται. Εμείς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καινούρια. Ε, τι γίνεται με τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώνουν παλιούς λογαριασμούς και μετά από τέσσερα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση με αυτή που ζούμε σήμερα. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα προκύψει και δεν μπορούμε να το δεχτούμε ελαφρά την καρδία. Και να το πούμε και στην αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να τα υπολογίσουμε πάρα πολύ ε, με μεγάλη ακρίβεια, αλλιώ εκείνοι που εκτελούν τα έργα και οι περιφέρειες έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Το έχω ζήσει και η ίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει στις περιφέρειες ότι ε, έχουν τρύπα χρηματοδότησης, αλλά ε, κατεβάζει διάφορες ιδέες για διάφορα δικαιολογητικά και έγγραφα που λείπουν για να καθυστερήσουν ε, τις πληρωμές και τους τρέχουν. Αυτό δεν αυξάνει την αποδοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής περιφέρειας. Γιατί είναι που είναι μεγάλη η γραφειοκρατία και αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν. Ε, θα πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής είναι ένα θετικό εργαλείο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα πρέπει να το προβάλλουμε και να το διαφημίζουμε στις περιφέρειες. Και δεν επιτρέπεται όταν έχουμε πρόβλημα στη χρηματοδότηση ή όταν έχουμε πολύ ψηλή ε, γραφειοκρατία να δυσκολεύουμε τους δικαιούχους και να μην τους πληρώνουμε με κάποιες παρελκυστικές ε, τακτικές. Επίσης έχει σημασία να λέμε ότι στην πολιτική συνοχής ε, δεν ζει κανείς μόνο από επιδόματα, επιδοτήσεις, αλλά υπάρχουν και χρηματοδοτικά μέσα αλλά είναι τόσο περίπλοκη η πρόσβαση σε αυτά που μπορεί να χρησιμοποιούνται λίγο, αλλά όχι αυτό που είχαμε φανταστεί όταν εκπονήσαμε το Γενικό Κανονισμό για τη Νέα Πολιτική Συναχής. Κάπου είδα το Γιάνν Όλμπριχτ, παρευρίσκεται. Και, ναι, με το Γιάννη είχα κάποιες επαφές για τα όσα έλεγε η Επιτροπή Προπολογισμών στη δική της έκθεση. Νομίζω γενικά συμφωνούμε, στην ίδια γραμμή κινούμαστε. Και πάλι έχουμε τη συζήτηση για τη διάρκεια ε, της ε, περίοδου της προγραμματικής των δημοσιονομικών προοπτικών και τα πολιτή πλαίσια και τα πολιτή προγράμματα όπως η πολιτική συνοχής ή ορίζον 2020 πόσο θα πρέπει να διαρκούν. Στην γνώμη μου λέω ότι η επταετής ε, προγραμματική περίοδος έχει επιτύχει στην πράξη. Ξέρω ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάθε φορά. Μπορώ να καταλάβω ότι καλό θα ήταν να προσαρμοστεί στη θητεία του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πενταετή η προγραμματική περίοδος. Αλλά για την πολιτικής συνοχής να κάνεις τέτοια φασαρία για πέντε χρόνια μέχρι να αρχίσει το σύστημα να τρέχει έχει περάσει πενταετία. Οπότε νομίζω ότι τα 7 έτη είναι μια καλή εμπειρία, ε, έχει δοκιμαστεί στην πράξη και έχει αποδώσει, αλλά διάβασα ότι η Επιτροπή Προπολογισμών σκέφτεται να... Ε, την ε, ετία, δηλαδή πενταετία και μετά άλλη μια πενταετία δεν ξέρω, δεν θέλω να προεξοφλήσω τίποτα και τα δύο είναι κάτι που θα μπορούσα να δεχτώ και να το συζητήσουμε τους σκιώδεις εισηγητές γιατί όχι. Τελικά όμως για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν, η συζήτηση δεν είναι ο χώρος που θα πρέπει να συζητήσουμε την πολιτική συνοχή και να παίξουμε αυτή την κολοκυθιά επταετία ή δύο φορές μία πενταετία. Δεν είναι η παρούσα γνωμοδότηση ε, το κατάλληλο σημείο για να γίνει αυτή η συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Αυτά πάρα πολύ σύντομα ε, τα ολίγα. Νομίζω και ελπίζω να συμφωνείτε και περιμένω τις προτάσεις σας για το πώς θα μπορέσω να βελτιώσω και να εμπλουτίσω την ε, όλη γνωμοδότηση. Θα κάνω, σας είπα, και προσωπικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, thank you very much. Now we open... Ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Νοβάκοφ, εκ μέρους του ΕΛΚΑ, πρώτος και ο Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Κρέτ, για την καλή γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία και για όλες τις συζητήσεις που είχαμε. Και τις τροπολογίες που είχα στο μυαλό μου. Η αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι πάντα μια κρίσιμη στιγμή για όλη την περίοδο προγραμματισμού, ιδίως όταν η περίοδο προγραμματισμού δεν είναι ακριβώ αυτό που περιμέναμε δυστυχώ το 2014-2020, αλλά θα είναι τελικά 2016-2020. Έχουμε τους κανόνες ε, νη 2 και νη σε διάφορα σημεία η γνωμοδότηση τονίζει τη σημασία των συνεργειών. Και δυστυχώς, παρότι η Επίτροπος Κρέτσου καταβάλει πολλές προσπάθειες, θα θέλαμε κάτι περισσότερο, ε, περισσότερη συνέργεια ανάμεσα στα ταμεία. Θα θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε κάνει στην αρχή για το σχέδιο Juncker, Είχαμε τα προγράμματα ΕΣΥΦ, των διορθωτικών δηλαδή και επενδυτικών ταμείων. Αλλά να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Το κοινωνικό ταμείο και το EGF, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, καλύπτουν το ίδιο θέμα και το κράτος μέλος επιλέγει ποιο από τα δύο θα χρησιμοποιήσει. Νομίζω ότι δημιουργεί γραφειοκρατία. και μπερδεύει τους ε, πιθανούς δικαιούχους. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτή την ε, αναθεώρηση ή αναπρογραμματισμό του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Λόγω των έκτακτων περιστάσεων που αντιμετωπίζουμε τώρα με τους πρόσφυγες, πρέπει να δούμε τι, θα κάνουμε. Ό,τι έχει περισσέψει από το παλιό, την παλιά περίοδο προγραμματισμού, καλό είναι να το χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τις χώρες που πλήττονται κυρίως από το προσφυγικό. Αλλά δεν θα πρέπει να το ξανακάνουμε στο μέλλον, γιατί δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση. Δεν θα τελειώσει το Ρώσο Νούμπο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει πάντως. Και δεν θέλω ό,τι έχουμε και, και δεν έχουμε να το ξοδέψουμε για να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό. Και να μας μένει τίποτα για τους νέους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους νέους επιχειρηματίες. Σας ευχαριστώ για την νομοδότησή σας ακόμα μια φορά και περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις τροπολογίες και πιστεύω ότι το έργο που θα προκύψει θα είναι πολύ καλό. Κύριο Λούερ, επόμενο συγκητή. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Κρέλ για αυτή την έκθεση που είναι ε, γενικά σωστή και ισορροπημένη. Πιστεύουμε ότι οι οροφές πληρωμών ε, του πολιτικού προγράμματος για την περιοχη 2010 2014-2020 θα πρέπει να τύχουν σεβασμού και δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν, δηλαδή ε, δεν υποστηρίζουμε αύξησή τους. Αντιθέτως, θέλουμε να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι, διαθέσιμοι πόροι. Η, μεταναστευτική κρίση, παρόλο ότι είναι τραγική, δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να αυξηθούν τα, οι οροφές. Η ομάδα μας τονίζει την σημασία ο προπολογισμό να είναι βιώσιμος ε, και να διατηρηθούν οι εξουσίες των κρατών μελών, ενώ θα πρέπει να εστιάσουμε πόρους σε συγκεκριμένα project ε, και να αποφύγουμε επικαλύψεις. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και καθυστερούμενες πληρωμές, όπως ε, που έχουν ήδη προκύψει στο, στην εφαρμογή του προγράμματος του, της περίοδου 2014-2020. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των πολιτικών συνοχής και να αποφύγουμε τις, τις ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες και γενικότερα στους δικαιούχους. Η, η αναφορά στα χρηματοπιστωτικά με εργαλεία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ε, επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτεί μόνο μέτρα που έχουν προστιθέμενη αξία. Εκεί που δηλαδή ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ρόλο που θα είναι πιο μεγάλος, πιο σημαντικός από το άθεσμα των εθνικών ρόλων, των ρόλων που παίζουν οι εθνικές διοικήσεις. Ε, επίσης δεν θα πρέπει να συνηθίσουν με ορισμένοι δικαιούχοι ε, να ξοδεύουν χρήματα ως αυτοσκοπό. Μετά, ο πολιετής προγραμματισμός έχει κάποια ε, ελαττώματα για το κρατικό μηχανισμό ε, γιατί στερεί ευελιξία αλλά ε, πάντοτε υπάρχει ένα θέμα ε, ισορροπίας ανάμεσα στην προβλεψιμότητα και στην ευελιξία. Θέλουμε την ευελιξία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το να αποφύγουμε η εμπροστοβαρής δαπάνη ποσό να μην οδηγήσει, να οδηγήσει σε ε, αύξηση των, ε, του συνολικού ποσού. Επίσης ε, δεν θα πρέπει η απλοποίηση να οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας και κοιτάξτε την, το κάτω μέρος της σελίδας 3 ε, της έκθεσης Κομισιόν. Ε, ελπίζω ότι θα αποφευθεί αυτό. Επίσης η απλοποίηση καταρχήν θα πρέπει να ωφελεί τους ετούντες και ενδεχομένως και τα κράτη-μέλη. Όχι όμως ιδιαίτερος να ωφελεί την ίδια την Κομισιόν και το προσωπικό της. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ επόμενη σκιώδη συγγήτρια είμαι εγώ. Οπότε επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω στα βουλγαρικά τη γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Κρέλ την εισηγήτριά μας και να αναφέρω κατόπιν και μερικά, ένα-δύο έτσι, πολύ σημαντικά ζητήματα. Στα οποία πιστεύω ότι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση με την κυρία Κρέλ. Η αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, ε, την πολιτική συγκυρία, την ε, μεταναστευτική κρίση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις ε, ε, συνέπειες της οικονομικής κρίσης που εμπολείς ακόμα δεν είναι γνωστές. Ε, έχουν παρουσιαστεί ήδη καθυστερήσεις πληρωμές στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ε, γι' αυτό το λόγο είναι λίγο ή μάλλον αδύνατο να υπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα των πόρων που διατίθενται. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, καθυστερήσεις και να κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους που διαθέτουμε και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστούν οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να βελτιώσουμε την ε, αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής. Θα πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα σε έναν προπολογισμό που προσανατολίζεται στα αποτελέσματα αφενός και στην απλοποίηση των διαδικασιών από την άλλη. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για τη χρηστή διαχείριση, χωρίς όμως να κάνουμε τα προγράμματα διαχείρισης των πραγμάτων υπερβολικά περίπλοκη. Οι ε, προγράμματα που έχουν σχέση με την εδαφική συνεργασία θα μπορούσαν να διαβρινθούν για να περιλάβουν και το προσφυγικό. Επίσης, κάποια, ε, κάποιες ε, δωρεάν χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις δηλαδή, θα μπορούσαν να συνδυαστούν με το πρόγραμμα, το σχέδιο Juncker ε, και ε, έτσι να δημιουργήσουμε κίνητρα και για ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε έναν ανοιχτό μηχανισμό συντονισμού για να εξασφαλίσουμε τη λογική συνέπεια να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις και να εξασφαλίζουμε συνέργειες ανάμεσα στα ευρωπαϊκά, τα εθνικά κονδύλια, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει προτάσεις βελτίωση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου έτσι ώστε ε, να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή ενός σχετικά περιορισμένου ε, ως γνωστόν προπολογισμού. Χωρίς να αλλάξουμε τις προτεραιότητες, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα απλοποίησης εφαρμογής και προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή συνέργεια ανάμεσα στα διαδοτικά ταμεία και τα άλλα προγράμματα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να, εξασφα συνδυάσουμε πόρους και από άλλα εργαλεία. Τα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τρόπο σωστό ε, και εφαρμόζοντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο κ. Σόμερτζέ ε, ε, έχει το λόγο κανονικά, δεν, εδώ, τον βλέπω. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Κρέλ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάθεση ε, του σχεδίου γνωμοδότησης. Είναι πάρα πολύ καλή. Ε, ε, συμφωνούμε και εμείς σαν ομάδα και την υποστηρίζουμε, το είπατε κι εσείς πολύ σωστά τονίσατε τη γενική σημασία των διαφορετικών ταμείων και της πολιτικής συνοχής και ως προς τους στόχους για το 2020. Και η πρότασή σας για την προσφυγική κρίση, καλύτερη αξιοποίηση των διαθροτικών ταμείων μας βρίσκει σύμφωνους και το υποστηρίζουμε και εμείς και επαυξάνουμε για την πολιτική συνοχή και τα διασωτικά ταμεία έχουν τεράστια σημασία και είναι μεγάλη πρόκληση το προσφυγικό. Είναι πολύ μεγάλη σημασία και πολύ σημαντικό να το λέμε στην γνωμοδότηση. Κάτι που μας λείπει λίγο για μας είναι η προστασία του κλίματος και πώς μπορούν τα ταμεία αυτά και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, να βοηθήσουν. Αυτά τα έχει εκπονήσει και η Λουξεμβουριανή Προεδρία και υπάρχει και η δέσμευση το 20% του ευρωπαϊκού προπολογισμού να πηγαίνει στην προστασία του κλίματος και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και μετά από τους στόχους του COP21 και την εφαρμογή του. Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της πρόσβασης στα διορθωτικά ταμεία, εμείς κανονικά ε, θα θέλαμε να αλλάξει λίγο η διατύπωση. Προτείνουμε μια μικρή αλλαγή. Ε, αυτή τη στιγμή η γνωμοδότησή σας μιλάει μόνο για απλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, financial instruments, αλλά χρειάζεται και μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Ξέρετε ότι εμείς είμαστε κάπως επικριτικοί απέναντι σε αυτά, γιατί κατά την άποψή μας δεν έχει αποδειχθεί η μεγαλύτερη χρησιμότητα και αποδοτικότητά τους. Εμεί θέλουμε ενισχύσεις, επιδοτήσεις και δάνεια, κλασικά δηλαδή. Θα κάνουμε και τροπολογίες. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι και μια ε, ευκαιρία για να μην πω υποχρέωση να σκεφτούμε και παραπέρα και θα κάνουμε και μια τροπολογία για ε, το ΑΕΠ αλλά και επέκεινα του ΑΕΠ. Δηλαδή και πέρα από το καθάριστο εθνικό προϊόν ε, να έχουμε και άλλα κριτήρια για την εχώρηση των κονδυλίων. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε και προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία μαζί σας. Η κυρία Βάνα, η μόλις μίλησε. Κύριε Νταμάτο. Η συνεισφορά του Κοινοβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου είναι σημαντική και για την Επιτροπή Προπολογισμού και για την Επιτροπή Ρέτζη, τη δική μας. Εκτιμώ λοιπόν το σχέδιο νομοδότησης της κυρίας Κρέλ που μιλάει για τα πιο σημαντικά στοιχεία. Την ανάγκη βελτίωσης της συνέργειας και του συντονισμού ανάμεσα στα πέντε ταμεία και άλλα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την απλούστευση, για την επιτάχυνση της εφαρμογής της ε, πολιτικής συνοχής και για το πρόβλημα των καθυστερούμενων πληρωμών. Ειδικά καλή είναι η παράγραφο όπου αναφέρονται οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα, τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες, ούτω ώστε ε, να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες, ούτω ώστε να υποδεχθούν του ε, τούτε άσυλο και άλλου μετανάστες, να δώσουμε μία επιπλέον βοήθεια σε αυτά τα κράτη-μέλη και σε αυτές τις περιφέρειες βέβαια, όταν επανεξετάσουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Λοιπόν, κάτι που θέλω να πω τώρα και θα τα παρουσιάσω και σε τροπολογίε. Καταρχάς, για το σημείο που αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι επιδοτήσει θα πρέπει να είναι μια αποτελεσματική μορφή υποστήριξης πολλών τομέων παρέμβαση του δημόσιου τομέα. Αλλά και θα πρέπει να το δεχτεί και στην γνωμοδότηση, θα πρέπει να δοθούν ε, και άλλε αποδείξει, να γίνουν και άλλε μελέτε για να αποδείξουμε ότι αυτά είναι αποτελεσματικά σε κάποιους τομεί πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι η, το εκτιμώντα 53 ε, του κανονισμού που μιλά για του ε, κανόνε που αφορούν τον προπολογισμό τη Ένωση, λέει ότι τα δημοσιονομικά εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με βάση μια αξιολόγηση που θα γίνει εκ των προτέρων που θα δείχνει τη μεγάλη αποτελεσματικότητά τους για την υλοποίηση των στόχων που είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με άλλες μορφές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των επιδοτήσεων. Δεύτερον, το θέμα των συνεργειών ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και άλλων πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραίο. Ε, οι συνέργειε ανάμεσα στο ορίζοντα 2020 και στα διαφορετικά ταμεία, αλλά ένα σχόλιο όταν τα ίδια λεφτά του ορίζοντα 2020 και του μηχανισμού ε, ΕΣΥΦ δηλαδή χρησιμοποιούνται για την ε, χρηματοδότηση του σχεδίου Juncker, τι νόημα έχει. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση, συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που λέγεται. Επίσης όλοι μας στο ψήφισμα της Επιτροπής μας είχαμε, που εγκρίθηκε το φθινόπωρο, τα είχαμε πει αυτά. Η απλούστευση όλων των ε, μέτρων, ούτως ώστε η πολιτική συνοχή να γίνει πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μην ξεχνάμε την ανάγκη να διατηρήσουμε τους σωστούς ελέγχους ε, κατά των ε, λαθών και κατά των απατών. Επίσης, να προσθέσω, όπως λέει και η συγγήτρια, το άρθρο 2 του κανονισμού του Συμβουλίου που αναφέρεται σε μια παράγραφο, λέει ότι οι εθνικές ε, χρηματοδοτήσεις, αυτό το front loading, η προκαταβολή δηλαδή, δεν πρέπει να μειωθεί όταν αναθεωρηθεί το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε όμω και το άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού, το οποίο λέει ότι για να λάβουμε υπόψη την ειδική ειδικά δύσκολη κατάσταση κάποιων χωρών που πλήττονται από την κρίση, μπορεί να γίνουν ε, στατιστικές προσαρμογές ε, ύψους 4 δισεκατομμύριων ευρώ. Θα πρέπει να δούμε πώ θα εφαρμοστούν αυτά τα δύο άρθρα του κανονισμού. Για να καταλήξω. Εμείς θεωρούμε ότι όντως πρέπει να προωθήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική για τις επενδύσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε το, το σχέδιο συμφωνίας από τις, ε, το σύμφωνο σταθερότητα συγγνώμη, από τις ε, εθνικές επενδύσεις και τα ποσά που παίρνουμε από αυτό δηλαδή από τις εθνικές επενδύσεις. Ωραία. Θα περάσουμε στον κύριο Άλμπρεχτ που έχουμε την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Ε, είμαι και εισηγητής ε, ε, στην Επιτροπή Προπολογισμού για την αναθεώρηση του πολιτισμού συνομικού πλαισίου και αντικαταστάτης εδώ. Έχω κάποιες προτάσεις να κάνω. Το κείμενο του της, ε, του προσχεδίου της δικής μας έκθεσης, της δικής μας νομοδότησης, είναι έτοιμο ε, από την Επιτροπή Προπολογισμού και χωρίζεται σε τρία τμήματα, θα το δείτε. Στην συζήτηση εδώ είναι επίσης σαφές ότι αυτά τα τρία τμήματα είναι τα εξής και πρέπει να είναι τα εξής. Πρώτον, μια πραγματική αξιολόγηση αναθεώρηση και η Επιτροπή Ρέτζι μπορεί να ζητήσει και από την Επιτροπή Προπολογισμού και από την Κομισιόν να αναθεωρήσουν ε, την ε, πολιτική συνοχής όχι στην επόμενη έκθεση, αλλά σε συνδυασμό με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πριν τι προτάσει Κομισιόν. Δηλαδή, πριν την αναθεώρηση του πολιτού πλαισίου να, γίνει, να γίνουν προτάσει ε, ε, να υποβληθούν προτάσεις για την αναθεώρηση ε, της πολιτικής συνοχής. Αναθεώρηση σημαίνει τι συνέβη τα πρώτα χρόνια και τι πρέπει να συμβεί τα επόμενα. Οπότε η πρώτη, το πρώτο στάδιο είναι η αξιολόγηση του τι έγινε στο περίοδο 14-16. Δεύτερον, εσείς για το έγγραφο που θα προετοιμάσει η Κομισιόν και θα ψηφίσει το, κοινό, το Συμβούλιο οι προτάσεις μας δηλαδή για το τι θα πρέπει να αλλάξει αμέσως, αμέσως όχι στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό είναι η αναθεώρηση, μετά την αξιολόγηση λοιπόν αναθεώρηση. με βάση τη καινούργια κατάσταση, σημερινή συγκυρία κλπ. κλπ, κλπ. Χρειαζόμαστε για τα επόμενα χρόνια, 16 με 20, να κάνουμε τι εξή αλλαγέ. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα. Ε, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να αναθεωρηθεί. Για παράδειγμα, οι καθυστερούμενες πληρωμές για το 17, 18, 19 και 2020. Γιατί ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα για την πολιτική συνοχή. Το είπε η Κωνσταντσε. Ε, θα ξαναντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των καθυστερήσεων. Οπότε τι πρέπει να αναθεωρήσουμε. Και τρίτον, ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία θα φορούν τις νέες ε, δημοσιονομικές προοπτικές, τις επόμενες. Γιατί ε, είναι ευκαιρία να πούμε τι αφορά το δεύτερο κομμάτι της προγραμματικής περίοδου μέχρι το 2020 και τι αφορά την περίοδο μετά το 2020. Ορισμένες αλλαγές πρέπει να γίνουν τώρα, ορισμένες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν μετά το 2020. είναι διαφορετικό αυτά που προτείνουμε να αλλάξουν τώρα, διαφορετικά αυτά που πρέπει να προτείνουμε να αλλάξουν μετά το 2020. Τέλος, ε, στην δική μας έκθεση ε, θα περιλάβουμε την πρόταση πενταετούς προγραμματισμού. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, επίμαχο. Το, ε, ε, θα, ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο έτος ε, των δημοσιονομικών προοπτικών. Ε, έχουμε πενταετή προγραμματισμό. Είμαστε ήδη στο τρίτο έτος και είμαστε ακόμα στην αρχή. Οπότε εμείς θα προτείνουμε ναι γενικά για το πενταετές, αλλά σε συγκεκριμένες πολιτικές που χρειάζονται ε, μακρόπρόθεσμο προγραμματισμό να προβλέπουμε πέντε συν πέντε χρόνια και η αναθεώρηση, η αξιολόγηση αναθεώρηση να γίνεται στα πέντε χρόνια, όχι στα τρία. Βέβαια, το Συμβούλιο θα διαφωνήσει, μπορεί τελικά να καταλήξουμε στα 7 συνολικά, όχι πέντε συν πέντε, αλλά πέντε συν δύο, Ε, πάντως τα πέντε για ορισμένες πολιτικές, για την πολιτική συνοχής είναι ανεπαρκέστατο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 7, αν όχι 10. Και ασφαλώς θα πάρουμε υπόψη και τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαν Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι εξαιρετική η δουλειά της. Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι παράγραφο 2 του σχεδίου γνωμοδότησής σας γιατί πριν το 2017 δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ε, το αποτέλεσμα. Είναι πολύ νωρίς για να καταλήγουμε σε συμπεράσματα αυτής της πολιτικής. Ανησυχώ ε, για τα στοιχεία και τις ημερομηνίες για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, ιδιαίτερα γιατί θα είναι πολύ χαμηλή η απορρόφηση σε ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα και τα στοιχεία απολύτως ανεπαρκή. Δεύτερον, εγώ διαφωνώ με την εισήγητη. Δεν συμφωνώ με την παράγραφο 9 του σχεδίου γνωμοδότησής σας. Η προγραμματική περίοδος θα πρέπει να είναι πενταετής. Άκουσα μόλις τον κύριο Όλμπριχτ Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι εάν προσαρμόσουμε την ε, προγραμματική περίοδο με την πολιτική θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε θα αυξήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα και τη λογοδοσία. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι έτσι προαιρετικό είναι στη διακριτική μας ευχέρεια, θα πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε μια εντολή συγκεκριμένη και έχει νόημα να συνδέσουμε και να προσαρμόσουμε ε, τη θητεία μας και την εντολή μας με την οικονομική ε, προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόν, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Την εισηγήτρια. Δίνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς η απλούστευση. Πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στην απλούστευση μετά τις συστάσεις της ομάδου. Θα χρειαστεί πολύς χρόνο ή θα το κάνουμε γρήγορα. Φυσικά υπάρχει το πρόβλημα του προπολογισμού. Υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιε γραμμέ προπολογισμού σημαντικέ, πρέπει να τι δούμε. Ε, βέβαια είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να αποφασίσουμε τι πρέπει να αλλάξει γιατί τα πράγματα είναι σε αρχική φάση. Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη την πρικοδότησή τους από τα διαρθρωτικά ταμεία και είναι δύσκολο να αλλάξουμε τα ποσά αυτά. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Κάποια άλλα πράγματα, ε, οι καθυστερούμενες πληρωμές, στο τέλος οι καθυστερούμενες πληρωμές θα είναι κάτι του, 2, του ύψους του 2 δις σχετικά μειωμένε, αλλά μπορεί να ξανα, ξαναυξηθούν μετά οι καθυστερούμενε πληρωμέ. Ε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, να τον αναγνωρίσουμε. Κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για τον προπολογισμό ε, όταν η Κομισιόν, Κομισιόν και το Συμβούλιο από την άλλη και από την άλλη η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο α, όταν συζητάνε τον προπολογισμό πάντα μιλάνε ε, για τις καθυστερούμενες πληρωμές. Ε, κάτι πρέπει να κάνουμε γιατί αλλιώς μέχρι το 2020 θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Επίσης, τι θα γίνει. Πότε θα κάνουμε κάποια πράγματα, θα τα κάνουμε νωρίς ή αργά στην περίοδο προγραμματισμού. Κάτι καινούργιο που θα ήθελα να πω είναι το αποθεματικό με βάση τις επιδόσεις. Ε, στο παρελθόν είχαμε αντιταχθεί. Θεωρούσαμε ότι είναι περιτό. Τώρα αυτά τα ποσά όμως, ε, στο τέλο περίπου περίοδου προγραμματισμού, τα ποσά από αυτό το αποθεματικό θα, θα δοθούν. Θα, ξανα, θα αλλάξουν τα ποσά και πότε θα δοθούν αυτά τα ποσά. Γιατί αυτό ε, θα επηρεάσει τον ετήσιο προπολογισμό και το τρέχον ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν το έχουμε πει αυτό, θα πρέπει να το συζητήσουμε και να το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρέσο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Κρέλα για τη γνωμοδότηση που είναι πολύ σημαντική γιατί προφανώς η, Επιτροπή Μπάτζ έχει αρμοδιότητα για τον προϋπολογισμό γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την, το ποσοστό του προϋπολογισμού που αφορά την πολιτική συνοχή που είναι σημαντική συνιστόσα. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική η γραμμή αυτή που αφορά το Ταμείο Συνοχής και για τη δική μας Επιτροπή. Δεύτερο. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, πραγματική και πλήρης αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, όχι μόνο μια αξιολόγηση. Γιατί όπως είπε και ο Όλμπριχτ, υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα πολύ σοβαρά εντός του προϋπολογισμού το θέμα των καθυστερούμενων πληρωμών. Αλλά το γεγονός ότι μονίμως το Συμβούλιο παίρνει σημαντικότατες αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις οικονομικές, χωρίς όμως ποτέ να αλλάξει τον προπολογισμό. Επομένως υπάρχει κίνδυνος η πολιτική συνοχής που σε αυτή τη φάση έχει καθυστερήσει λόγω της καθυστερημένης απόφασης που ελήφθη για το Πουδουδού και επομένως και για το προϋπολογισμό και θεωρείται ανεπαρκής. Εάν θέλετε λοιπόν να πάρετε ακόμα περισσότερους πόρους από την πολιτική συνοχή για να τα πάτε αλλού αυτά τα λεφτά, ε, υπάρχει πρόβλημα. Επίσης θα συσσωρευτεί καθυστέρηση. Και εξαιτία αυτής της καθυστέρησης ε, θα, μειωθεί το, θα μειωθούν οι, ε, οι δεσμεύσεις πληρωμών. Η συγγνώμη. Επομένως, η ενδιάμεση αναθεώρηση ε, της, ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε αν όλη η δουλειά που κάνουμε, που κάνει η Επιτροπή μας, που κάνει η Κομισιόν, που κάνει η Επίτροπος και δουλειά την οποία εμείς ελέγχουμε για την απλούστευση, αν γίνεται σωστά και αν είναι σημαντική. Γιατί αλλιώς μπορεί από, από το, την πολιτική συνοχής να αφαιρεθούν πόροι. Κι όμως, οι πόροι είναι όλο και πιο απαραίτητοι για τους ε, τοπικούς φορείς και τις περιφέρειες για να κάνουν αναπτυξιακή πολιτική. Αλλά λόγω των περιπλοκών, λόγω των καθυστερήσεων, τελικά είναι πολύ, έρχονται πολύ αργά αυτοί οι πόροι και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα, το αν θα έχουμε 7 αιτία ή 5 σε 5 χρόνια, αυτό το θέμα συνδέεται πάρα πολύ με το προηγούμενο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γενική πολιτική προπολογισμού της Ένωσης, τη δημοσιονομική πολιτική, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η κοινοβουλευτική θητεία και η περίοδος προγραμματισμού να είναι το ίδιο πράγμα, πέντε χρόνια δηλαδή. Αλλά έτσι όπως έχει σήμερα η πολιτική συνοχής ε, μέσα σε πέντε χρόνια δεν μπορεί να δώσει καρπούς. Έτσι, δεν φτάνουν τα πέντε χρόνια. Υπάρχει το εξή πρόβλημα. Το 5 συν 5 καταρχά να το έχουμε για την πολιτική συνοχή, αλλά αυτό να μην σημαίνει μία περαιτέρω επιμήκυνση των χρόνων, α πούμε. Ε, δηλαδή, ακόμα περισσότερο χρόνο και ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση για να εκταμιευθούν τα ποσά. Αλλά τέλο πάντων, αυτό θα το συζητήσουμε όταν μιλήσουμε για την αναθεώρηση τη πολιτική συνοχή. Τώρα για το θέμα μα. Εγώ νομίζω ότι Πρέπει να δούμε λιγάκι αυτό το θέμα των χρόνων, δηλαδή. Πόσα χρόνια, 7 ή 5 συν 5. Γιατί από τη μία τα λεφτά πρέπει να ξοδευτούν όλα. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνουν οι εκταμιεύσει αυτέ με τρόπο τρομερά αργό. Γιατί ο χρόνο κυλάει πολύ, πάρα πολύ γρήγορα, οι οικονομικέ συνθήκε αλλάζουν έτσι άρδιν και πολύ γρήγορα. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο να επιμηκύνουμε ακόμα περισσότερο το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο χρειάζεται που χρειαζόμαστε για να δαπανίσουμε τα ποσά της πολιτικής συνοχής, αυτό είναι περιττό. Επίσης, το πρόβλημα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Καλό είναι οι δεσμεύσει και οι πληρωμές να έχουν μια συνέπεια, έτσι. Γιατί όταν καθυστερούμε και δεν εκταμιεύουμε, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τρομερές ε, καθυστερήσεις στις πληρωμές ε, στη δεύτερη φάση, εάν καθυστερήσουμε το... την εκταμίευση στην πρώτη φάση. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα των καθυστερούμενων πληρωμών. Πρέπει να το θέσουμε με έμφαση. Είναι από τα προβλήματα που δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις μετέπειτα φάσεις ε, της περίοδου προγραμματισμού και στη διαχείριση των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Και τις ε, δυσκολίες αυτές ποιος τις έχει, οι περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση βέβαια. Κύριο Σχέτμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Το προσχέδιο είναι πολύ καλό. Καλύπτει τα πιο σημαντικά ζητήματα. Αλλά θα ήθελα να δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση, να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να εξεταστεί η πολιτική συνοχής για μετά το 2020. Η πολιτική συνοχή ε, θα πρέπει να διατηρηθεί με επαρκή χρηματοδότηση ως αν αυτόνομη πολιτική και στην περίοδο μετά το 2020. Χαίρομαι που κάνει λόγο εισηγήτρια για τις συνέργειες ανάμεσα στα διάφορα διευθυντικά ταμεία, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε να πάμε λίγο πιο μακριά γιατί οι εκκλήσεις για συνέργειες έχουν πολλαπλασιαστεί αλλά αυτό δεν έχει δώσει καρπούς μέχρι τώρα. Οι εκκλήσεις δηλαδή δεν έχουν μεταφραστεί σε πράξη επαρκώς. Θα πρέπει ε, να ζητήσουμε συνέργειες ανάμεσα στο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αλλά να μην μείνουμε στις εκκλήσεις, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να το προωθήσουμε. Γιατί οι συνέργειες στην πράξη είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Ας είμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι. Ας περιοριστούμε στις συνέργειες μεταξύ Κοινωνικού Ταμείου και Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Επίσης χρειαζόμαστε 7 ετή περίοδο, προγραμματική περίοδο. Και αυτό γίνεται εμφανές από το πόσο αργά προχωρούν τα προγράμματα και πόσο μικρή είναι αυτή η περίοδος η πενταετής αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Κύριε Σπόλτσακ, ευχαριστώ πολύ ε, για ε, το θέμα αυτό θα ήθελα να πω τα εξής δύο για την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Κρέλ θέτει αυτό το ζήτημα και το αναφέρει και στην γνωμοδότησή της, συγκεκριμένα στην παράγραφο υπαριθμό 7, όπου ακριβώς αναφέρεται στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και εκείνους που ζητούν άσυλο. Πραγματικά εγώ θα μιλούσα εδώ για πολιτική μεταναστευτική και πολιτική ασύλου και θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε αυτά τα πράγματα γιατί δεν είναι τα ίδια τα κράτη εκείνα που υποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες θα πρέπει να έχουν και οικονομική υποστήριξη. Συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε και να περιγράψουμε πώς θα κατανέμονται αυτά τα κονδύλια και ποιος θα είναι ο μηχανισμός. Και μετά, για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς και τις καθυστερημένες πληρωμές αναφέρθηκε η κυρία Μπρέσο σε αυτό. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική συνοχής μόνο. Είναι πολύ ευρύτερο και πολύ σοβαρότερο. Θα πρέπει να το καταδικάσουμε, διότι εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ήταν ε, στη συζήτηση ο κύριος Πόλτσακ και θα δώσω το λόγο ε, στην κυρία Ρουπιάνη από τη Γενική Διεύθυνση ε, Στον κύριο Ρουπιάνη, συγγνώμη. Θα είμαι σύντομος, κυρίως επειδή συμφωνούμε με τις βασικές αρχές του προσχεδίου γνωμοδότησης. Αυτές αντικατοπτρίζουν και τις δικές μας απόψεις σε ό,τι αφορά τα διαθροτικά και επενδυτικά ταμεία και τη σχέση τους με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την αθεώρησή του. Για μας ε, πρώτη προτεραιότητα είναι η απλοποίηση κάτι το οποίο ζητήσατε κι εσείς. Ε, θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις ε, της ε, Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου. Δεύτερη προτεραιότητα, να εστιάσουμε περισσότερο στα αποτελέσματα, Παρόλο την πρόοδο που έχει ήδη γίνει, ε, σχέση με την ε, των με την ευθυγράμμιση με τα αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, τρίτον, η πολιτική μας να είναι πιο ευέλικτη και να μπορεί να προσαρμόζεται στις καινούριες προκλήσεις χωρίς να αλλάζουμε τη δομή της. Αυτή είναι η τρίτη προτεραιότητα, πολύ σημαντική για την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την παραφορά 4, ε, εν παραλίλω με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα γίνει και η τεχνική προσαρμογή. Δηλαδή θα αναθεωρήσουμε τις σπόρους που πηγαίνουν στα κράτη-μέλη, ε, τους πόρους μάλλον τους εθνικούς σπόρους σε σχέση, ε, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε. Έτσι ώστε να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά για την πολιτική συνοχή ε, και για την περίοδο 2017-2020. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό το προβλέπει το άρθρο 92 του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων και το άρθρο 7 του Κανονισμού για το Πολιωτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Τέλος, όχι άμεσα σχετιζόμενο με την αναθεώρηση, αλλά κάτι παράλληλο, θα είναι η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων οι οποίες λίγουν. Η, το top-up, ε, δηλαδή το ποσοστό συγχρηματοδότησης που έχει αυξηθεί για χώρες οι οποίες βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και η απόφαση για το να παραταθεί αυτός ο ειδικό συντελεστής συγχρηματοδότησης για την Κύπρο. Ευχαριστώ κύριε Φανλίστερ Ρόι, ζητώ συγγνώμη, έχετε το λόγο. Μήπως δεν σήκωσα το χέρι μου αρκετά ψηλά, ξέρω εγώ πώς να με βλέπατε. Σύντομα, ε, για να μην παρατείνω τη συζήτηση. Είναι πολύ καλή αυτή η βάση ε, για να εργαστούμε επί του κειμένου και να εκθέσουμε και να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας. Προσωπικά, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά θα πρέπει να εξηγούμε ξανά και ξανά τι κάναμε στους νέους κανονισμούς για την ε, κατάσταση, τη θεματική, για τις νέες πολιτικές, για τα αποτελέσματα, για το πώς συμμετέχουν οι διάφοροι εταίροι. Κάθε φορά πρέπει να τα εξηγούμε αυτά. Είναι πάρα πολύ λογικά ότι πρέπει να έχουν αποτελέσματα ε, το 2017 οι προσπάθειές μας. Με αυτό έχουμε αποφασίσει στο κάτω-κάτω. Ας φροντίσουμε να γίνει. Και αν υπάρξει ανάγκη αναθεώρησης, ε, αναπροσαρμογής, ξέρω εγώ, και για νέα αποτελέσματα, για νέες προτάσεις, ας δούμε πρώτα τα αποτελέσματα, γιατί να προτείνουμε εκ των προτέρων. Και πάλι θα πρέπει να τα εξηγήσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται μια μακρύτερη περίοδος. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό. Ε, τα έχουμε αποφασίσει ήδη. Και θα πρέπει να τα λέμε ξανά στη συζήτηση ε, τα διαφορά ε, θέματα και τις διάφορες ενότητες. Στο σημείο 4 λέτε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο προπολογισμό. Και ακούσαμε καλά νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αυξηθεί κιόλα. Όχι μόνο δεν θα περικοπεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν μερικοί θεωρούν ότι μέχρι το 2020 θα αλλάξουν τον προπολογισμό, θα αλλάξουν την πολιτική μάλλον και θα βάλουν αμέσω χέρι στον προπολογισμό, πλανώνται. Καλό είναι που το είπε και ο κύριο Βόν το είπε. Το αποθεματικό για τις επιδόσεις. Και εγώ όσο γίνεται θέλω να αξιοποιηθεί αυτό, αλλά να δούμε ποια κατάσταση έχουμε. Είναι για μετά το 2020, είναι στα δικά μας χέρια. Πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, πώς μπορούμε να αντλήσουμε από εκεί η χρηματοδότηση στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και τελευταίο σχόλιο. Με το τι αναμένουμε ε, σε σχέση με τις υπερήμενες πληρωμές. Αν έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταθέσει ένα πρόγραμμα δράσης αρκετά αποτελεσματικό για την παλιά περίοδο, έχει καλός. Η μόνη ερώτηση είναι τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τις καθυστερείς πληρωμές και διδαχτήκαμε τίποτα από όλα αυτά. Τι θα κάνουμε στο μέλλον. Είναι μοναδική ευκαιρία που έχει η Επιτροπή μας Περιφερειακής Ανάπτυξης να αναπτύξει ακριβώς και να προβάλλει τις θέσεις της. Και να δούμε τι θα γίνει την επόμενη διετία στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. now... Ευχαριστώ. Κυρία Κρέλ. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά ε, όλους σας και τους συναδέλφους για τις προτάσεις. Να επαναλάβω μερικά σημεία. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή μας Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι επιφυλακτική και να μην ζητήσει αύξηση των μέσων με την αναθεώρηση και με τη νέα προγραμματική περίοδο. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Τώρα αυτό δεν είναι του παρόντος. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να διαπληκτιζόμαστε για το τι προπολογισμό θα επιθυμούσαμε. Ειλικρινά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλο περιθώριο ελιγμών και χειρισμών, εκπείρασα το λέω αυτό. Πάντως αυτό που θα πρέπει τώρα να αγωνιστούμε είναι να μην μα αφαιρέσουν τίποτα, όχι να αυξηθεί ο προπολογισμό. Γιατί υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα που καραδοκούν να μα βάλουν χέρι στα λεφτά και στον προπολογισμό τη πολιτική συνοχής και να τον περικόψουν. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε και πάλι το εξή. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω ούτε τους εθνικού ε, προπολογισμού, μάλλον τι αναλογεί σε κάθε χώρα, ε, ούτε ζητώ επιπλέον κονδύλια για το προσφυγικό. Υπάρχει όμως μια ευελιξία στα 4 δισεκατομμύρια που σας είπα, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει ένα περιθώριο και μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε με ευφύ τρόπο. Δεν ξέρω, ορισμένες χώρες αν έχουν αλλάξει με βάση τους νέους, τους δείκτες κτλ. Να δούμε αν υπάρχουν υπόλοιπα leftovers ε, που να τα μεταφέρουμε εκεί. Και βέβαια η πολιτική συνοχή δεν, είναι πρωταρχικ... δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο να λύσει το προσφυγικό, το μεταναστευτικό ή το θέμα του ασύλου. Προφανώς δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά η ένταξη κάποιων ανθρώπων ή εκείνων που έχουν ζητήσει άσυλο ή που μπορεί να είναι και μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από σήμερα είναι στόχος ε, μεταξύ των στόχων της πολιτικής ε, συνοχής. Δεν είναι αποκλειστικός, αλλά προβλέπεται ήδη σήμερα. Οπότε καλό θα ήταν χωρίς να αλλάξουν οι προπολογισμοί, αλλά μπορεί να αλλάξει το ΕΣΠΑ, ας πούμε, κάθε χώρα και να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από εκεί για τους πρόσφυγες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε, ας πούμε, να το αποφύγουμε. Ούτε θα χαθεί αυτό αν σταματήσουν να έρχονται πρόσφυγες, γιατί είναι παρόντες αυτοί που έχουν ήδη φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ένταξή τους στην κοινωνία είναι μια διαδικασία χρονοβόρα που θα χρειαστεί πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το προσωρινό. Το είδαμε και τους τελευταίους μήνες και τον τελευταίο χρόνο. Και στο παρελθόν θα πρέπει να ε, ανατρέξουμε σε δεκαετίες ολόκληρες. Εδώ μιλάμε ακόμα για μετανάστες της δεύτερης και της τρίτης γενιάς που ζουν στα κράτη-μέλη και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ε, καταστάσεις. Η αναθεώρηση της πολιτικής θα πρέπει να συμβαδίζει και με την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει δίκιο ο Γιάνν Ολμπριχτ. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε για κάποια αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε τι έχει γίνει ήδη μια αξιολόγηση των ε, προγραμμάτων, των έργων της πολιτικής συνοχής, της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Αν δεν ξέρουμε τι κάνουμε, ε, ή τουλάχιστον να έχουμε κάποιες ενδείξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι συμβαίνει, πώς να αναθεωρήσουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πώς να κάνουμε προτάσεις για μελλοντικές αλλαγές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με μεγάλη χαρά να τα ξαναδούμε και να τα συζητήσουμε και να τα βάλω και στη γνωμοδότησή μου γιατί πρέπει να γίνει. Κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό είναι να κοιτάξουμε ποια είναι ε, η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Αλλά νομίζω ότι έχουμε έξτρα έκθεση ξεχωριστή στην Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να μπει στη δική μου γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμών. Πολλό δε μάλλον που το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης δεν είναι τμήμα του, ε, ε, δικού μας προπολογισμού της πολιτικής συνοχής. Αλλά είναι εικονικά ένα στοιχείο τμήμα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να έχει παρόμοιους στόχους με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά είναι ανεξάρτητο από την πολιτική συνοχή. Θα μπορούσαμε να το εντάξουμε εδώ, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Συμφωνούμε λοιπόν απολύτως για την απλοποίηση, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, καμία αντίρρηση. Και επίση συμφωνούμε για τη συνέργεια και φοβούμε ότι το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες και με τον ορίζοντα 2020 θα έρθουμε να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι οι συνέργειες αυτές που θα επιθυμούσαμε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και πάλι. Όπως και το θέμα του backlog των καθυστερήσεων σπληρωμές να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει προτάσεις για το πώς φαντάζεται να απορροφηθεί. Γιατί δεν μου, αρκούν, δεν αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα, το αποθεματικό των επιδόσεων, το performance reserve, ε, το Κοινοβούλιο είπε ότι έτσι όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαπραγματεύτηκε μαζί μας, ε, δεν είναι ουσιαστικό αποθεματικό επιδόσεων, αλλά κανονικά ο στόχος θα ήταν να επιβραβεύονται τα καλά έργα, οι καλές περιφέρειες ε, και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι ότι έχει μοιραστεί ήδη αυτό το αποθεματικό στα διάφορα κράτη και οι κατευθυντήριες γραμμές για το πώς χρησιμοποιούνται και το κατόφλι είναι τόσο χαμηλό που θα πρέπει να είσαι ουσιαστικά ανόητος για να μην επωφεληθείς από εκεί και δεν είναι κανένα ουσιαστικό ε, απόθεμα επιδόσεων. Και όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Είτε στο μέλλον θα οργανώσουμε ε, στην πολιτική συνοχή με τέτοιο τρόπο την ευελιξία μας για να μπορούμε να αντιδρούμε σε συγκεκριμένες προκλήσεις, ναι, περιστάσεις, κρίσεις, απρόβλεπτα και απρόπτα, κάθε είδους, είτε θα ε, κάνουμε ένα ουσιαστικό αποθεματικό για τις επιδόσεις, το οποίο δεν θα μπορούμε να μοιράζουμε εκ των προτέρων. Αυτό στην αναθεώρηση της πολιτικής ενοχής πρέπει να συζητηθεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να το αλλάξουμε εμείς. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο διατηρώ αμφιβολίες σχετικά. Γιατί κανονικά και ο γενικός κανονισμός θα πρέπει να αλλάξει με όλη τη διαδικασία που συνεπάγεται. Και θα πάρουμε λεφτά από τα κράτη. Να δω το κράτος μέλος που θα γυρίσει λεφτά. Οπότε με το Συμβούλιο αποκλείεται να τα βρούμε. Αλλά για τη μελλοντική πολιτική ε, συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης, η σύνδεση της συνέργειας και το δικαίου ε, των κρατικών ενισχύσεων, στο οποίο αναφερθήκατε εσείς, Πρόεδρε, έχει σημασία να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Πολλά πράγματα δυσκολεύουν τη ζωή μας γιατί το δίκαιο περί ενισχύσεων δεν συνάδει πολλές φορές ε, με αυτά που κάνουμε στις διάφορες κατηγορίες στην πολιτική συνοχή. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Να υπάρξει καλύτερο συντονισμός των στόχων των, ε, του δικαίου κρατικών ενισχύσεων από τη μια και τη συνοχή από την άλλη. Τώρα το θέμα της πενταετίας ή επταετίας. Κύριε Χέτμαρκ Να είστε βέβαια στην περασμένη φορά που το συζητήσαμε αυτό το θέμα, δεν μας πήρε μόνο μέρες, αλλά εβδομάδες και μήνες ολόκληρους, αν θυμάμαι καλά. Είναι πολλά τα επιχειρήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Απλώς να πω το εξής. Και έχει απολύτως δίκιο ο Γιάννη Όλμπρεχτ για την πολιτική συνοχής είναι αδύνατο να είναι η περίοδος λιγότερη από 7 χρόνια. Δεν αξίζει τον κόπο όλη αυτή η ιστορία και οι μπελάδες. Και αν έρχεστε και μου λέτε πενταετία τώρα για την προγραμματική περίοδο για την πολιτική συνοχή, αυτό σημαίνει κατάργηση της πολιτικής. Κάτι άλλο όμως που θεωρώ χρήσιμο είναι να συζητήσουμε αυτό το δύο φορές πέντε χρόνια. 5 συν Όντω, μετά την πρώτη πενταετία μπορεί κανεί μια ουσιαστική αναθεώρηση πολιτική συνοχή ή αξιολόγηση και μετά να σκεφτούμε αν αυτή η ευελιξία συμπεριληφθεί, αν μπορεί να αλλάξει κάτι μετά την πενταετία χωρίς να προκληθεί σάλος και κατακραυγή από τα κράτη-μέλη κάτω τα χέρια από τα λεφτά μας. Και τώρα η επταετία μπορεί να είναι όντως μεγάλο διάστημα γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα ισχύει και τι θα επικρατεί το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία μια στοιχειώδης ευελιξία. Και εξού και αυτή η κατασκευή ή η σκέψη 5 συν 5 είναι καλό. Και αντί για μία περίοδος επτά Αλλά αν είναι μία περίοδος πέντε ετής και τίποτα άλλο, έτσι και, και το, βγείτε και το πείτε σε κανένα δήμαρχο, περιφερειάρχη, κοινοτάρχη ή πρωθυπουργό, θα σας αποπάρουν. Αλλά αυτά τα πέντε συν πέντε χρόνια είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ως ιδέα και αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε. Που θα ασχοληθούμε στο μέλλον αυτή, δεν αμφιβάλλω. Απλώς τώρα θα πρέπει να το πούμε στη γνωμοδότηση με αυτόν τον τρόπο. Εγώ το αφήνω έτσι κάπως αόριστο, ότι αυτή η πιο μακροχρόνια περίοδος ε, αποδείχθηκε στην πράξη χρήσιμη, χωρίς να κάνω προτάσεις για το μέλλον. Δεν ξέρω, αν βρούμε κάποια άλλη διατύπωση, έχει θαλός. Λιγότερο από 7 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην πράξη δεν εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα. Αυτά νομίζω με ότι κάλυψα και απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Καλά, θα τα ξαναπούμε. Περιμένω τις τροπολογίες σας και έχουμε και τούτη τη βδομάδα συνεδρία των σκιωδών εισηγητών για να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε για κοινού συμβιβασμούς και προτάσεις. Δεν νομίζω είναι δραματικά τα πράγματα. Συμφωνούμε στη γενική κατεύθυνση πάνω κάτω όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για τις οπολογίες. 21 Απριλίου, 5η, 5 η ώρα το απόγευμα. Και τώρα, θα περάσουμε στην εδρία των συντονιστών. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη αναβάλλεται. Άρα περνάμε κατευθείαν στην εταιρεία των συντονιστών. Καλώ τους συναδέλφους που δεν είναι συντονιστές, παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Και κλείνει η τακτική συνεδρία της Επιτροπής μας.